Mes chers collègues, bonjour. Nous allons commencer nos travaux. Bonjour, Monsieur Lungril. <laughs> Καλή σας μέρα. Alors, vous... Καθίστε παρακαλώ. Δεν θα ζεσταθείτε σε αυτήν την αίθουσα γιατί έχουμε κλιματισμό. Επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε Σχέδιο ημερήσια διάταξη. Ε, ρωτώ ε, εάν μπορείτε να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Από ό,τι φαίνεται δεν έχετε αντιρρήσει. Έγκριση των πρακτικών τη 30η Μαου. Επίση, ε, εάν δεν υπάρχουν αντίθετε απόψει, μπορούν να εγκριθούν τα πρακτικά. Δεν έχω ιδιαίτερε ανακοινώσει να σα κάνω σήμερα. Επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά Σχετικά με το θέμα του, για το οποίο συντάκτρια είναι η κυρία Ζακλίν Φώστερ. Επομένως, Πρόκειται για ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, κυρία Φώστερ, αυτό το οποίο ε, σας απασχολεί ε, στην γνωμοδότησή σας, ταυτόχρονα και για το περιβάλλον ε, και για τις αεροπορικές δραστηριότητες. Οι σκιώδεις εισηγητές έχουν συναντηθεί ήδη, έχουν συζητήσει επί σειράς ε, συμβιβαστικών προτάσεων και επομένως θα σας δώσω το λόγο ε, κυρία Φώστερ και μετά θα δώσουμε το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές και φυσικά ε, και σε όποιον βουλευτή θέλει να εκφράσει άποψη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είναι αρκετά σφιχτό το πρόγραμμά μας, γι' αυτό σας λέω ε, εξ αρχής ότι κυρίως για τους, ε, ε, ε, για τους συναδέλφους που δεν είναι σκιώδεις συγητές, ο χρόνος αγόρευσής τους ε, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα με δύο λεπτά. Έχουμε και εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φαντάζομαι θα θελήσουν να πάρουν τον λόγο επί των θεμάτων που θα έχουν προκύψει και μετά θα ξαναδώσω εν τέλει τον λόγο στην κυρία Φώστερ για να ολοκληρώσει. Κυρία Φώστερ. Θα λοιπόν να ξεκινήσω ε, αναφερόμενοι σε ε, κάποιου συναδέλφου που δεν έχουν άμεση σχέση με την έκθεση. Και να του πω ότι αυτή η έκθεση έχει άμεση σχέση με την αναστολή τη απόφαση. Δηλαδή, προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ε, εκπομπών, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ευρωπαϊκό. Ένα ευρωπαϊκό που συστήθηκε πριν από κάποια χρόνια και δεν λειτουργήσε αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει αρκετή δουλειά και γι' αυτό λοιπόν και εγώ είμαι σε θέση να στηρίξω, ήμουνα σε θέση να στηρίξω την Επίτροπο Μπούλκο πέρυσι στο Μόντρεαλ στον Καναδά. Ο βασικός στόχος, όπως σας είπα, είναι να ανασταλεί η απόφαση. Γιατί αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι ένα παγκόσμιο σύστημα, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2021. Ως εκ τούτου, η δική μας ε, η αρμοδιότητα είναι να σταματήσουμε εκεί που βρισκόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουν οι διαπραγματευτές και δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τις άλλες 163 χώρες, να καταλήξουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο ελπίζουμε ότι θα ισχύει σε παγκόσμια εμβέλεια. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι ότι θα πρέπει να έχουμε κατακαιρματισμένα συστήματα, αλλά ένα σύστημα οικουμενικό και παγκόσμιο. Και το ευχάριστο είναι ότι πρόκειται για ένα προαιρετικό σύστημα, αλλά από τη στιγμή που έχουν υπογράψει οι χώρε, τότε πια δεν είναι προαιρετικό το σύστημα. 70 χώρε έχουν υπογράψει, οι οποίε βεβαίω ε, του αντιστοιχεί το 85% των ε, εκπομπών. Μέχρι εκεί λοιπόν είναι ευχάριστα τα νέα. Ας πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, γιατί σας είπα ότι όλοι επιθυμούμε να επιτευχθεί αυτό το παγκόσμιο σύστημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδης ηγητές, γιατί εκτός από τους συντονιστές προσπάθησαν να ενισχύσουν τη θέση μας ε, όσον αφορά τις συζητήσεις για αυτή την αναστολή της απόφασης και τη σχετική νομοθεσία. Ε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, εκεί δεν τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια θετική, ε, μια δική μας ισχυρή θέση στον τριμερή διάλογο. Στο Στρασβούργο αυτό που μπόρεσα να κάνω είναι να επιτύχω αρκετούς συμβασμούς και μπόρεσα λοιπόν να λάβω υπόψη μου όλες τις προτάσεις του ΕΛ και των Σοσιαλδημοκρατών των Φιλελευθέρων και φοβάμαι μόνο μία ή δύο τροπολογίες των ε, συναδέλφων μας ε, από ε, την ομάδα των Πρασίνων και την ομάδα της ΓΚΟΕ. Εξάλλου υπάρχουν και κάποιοι σοσιαλιστές οι οποίοι είχαν περίπου τις ίδιες τροπολογίες όπως και οι πράσινοι και δυστυχώς αυτές οι τροπολογίες επί των οποίων θα ψηφίσουμε αύριο δυστυχώς αυτές δεν είναι συμβατές με την κατεύθυνση που πρέπει να αναλάβει η ε, έκθεση. Να ήθελα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάτι, ότι ε, για πρώτη και για δεύτερη φορά όσον αφορά την αναστολή της απόφασης υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στους σοσιαλιστές, ε, το ΕΛΚ, τους φιλελεύθερους, το ECR και κάποια άλλα μεμονωμένα μέλη, γιατί νομίζω ότι όλοι μας συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατότητα για κάτι που το θέλουμε σε παγκόσμια εμβέλεια. Θέλω τώρα να αναφερθώ σε τρεις τομείς δεν θα μπω σε συμβαστικές προτάσεις. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία τώρα είναι να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν δύο προγράμματα το παλιό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρί ε, ανταλλαγής εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το σύστημα της ε, ανταλλαγής εκπομπών ήθελε να ορίσει συγκεκριμένα όρια. Το νέο το παγκόσμιο σύστημα, το σύστημα Κορσία όπως αναφέρεται, θα είναι ένα σύστημα αντιστάθμισης των εκπομπών και βλέπετε λοιπόν ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο γραμμικό Εγώ δεν συμφωνώ γιατί αυτός ο γραμμικός παράγοντας ε, κατ' ουσίαν έχει σχέση με το παλαιότερο σύστημα και ο γραμμικός παράγοντας δεν ταιριάζει στο νέο σύστημα. Αυτά ε, τουλάχιστον έτσι εγώ αυτό έχω να προτείνω. Επίσης πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε επικάλυψη, ε, δεν μπορεί να υπάρχει σύγκρουση με αυτά που θα κάνουμε στο μέλλον, γιατί από τη στιγμή που θα έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα, κατά την άποψή μας, τη δική μου τουλάχιστον, αυτό το παγκόσμιο σύστημα θα πρέπει να ισχύει και για πτήσεις από τρίτες χώρες, αλλά και για ένδοενωσιακές πτήσεις. Γιατί μια πτήση μεταξύ και Παρισίου είναι μια μια διεθνή πτήση και έτσι πρέπει να ισχύει και εκεί η νέα μας πρόταση. Το γεγονός όμως ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα κράτος μέλος ή από μια εταιρεία να λειτουργούν διαφορετικά προγράμματα, θα πρέπει το ίδιο πρόγραμμα να ισχύει και για τις εσωτερικές πτήσεις. Άρα δηλαδή αυτό το έχουμε συμπεριλάβει σε μια συμβαστική πρόταση. Όσον αφορά κάποια άλλα βασικά θέματα, στο αρχικό πρόγραμμα όταν ε, συγκεντρώναμε πόρους, νομίζω ήταν απόλυτα ασαφές ε, γιατί επρόκειτο για πόρους που προέκυπταν από τις ε, εκπομπές, από την αεροπλοεία. Ε, υπήρχαν κάποια προγράμματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Εμάς όμως δεν μας αρέσει αυτό, γιατί το θέμα είναι ότι αν αυτά ισχύουν για την αεροπλοεία και τον αεροδιαστημικό κλάδο υπάρχουν σχετικά προγράμματα, ο καθαρός ουρανός 1, ο καθαρός ουρανός 2. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια ε, τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί στην έρευνα και την τεχνολογία. Έχουμε τον ενιαίο ουρανό, έχουμε όλα αυτά τα προγράμματα αλλά και μελλοντικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να περιοριστούν ε, οι εκπομπές. Μιλάμε τώρα για ένα σχετικό πρόγραμμα ε, με περιορισμού διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα κράτη-μέλη να έχουν πόρους από το παγκόσμιο σύστημα και αυτά, αυτούς τους πόρους θα τους επενδύσουν σε έρευνα και τεχνολογία που θα οδηγήσουν στο να περιοριστούν εκπομπές από την αεροπλογία και τον αεροδιαστημικό τομέα. Αυτά όσον αφορά την κατοχήρωση των πόρων. Υπάρχει και κάτι άλλο, νομίζω είναι η τροπολογία υπερθμών 70. Εκεί επαναλαμβάνουμε ε, το... Ε, αυτό που έχουμε πει και στην αρχή, δοκιμαστικές πτήσεις, ε, διπλωματικές ε, πτήσεις, ε, εκπαιδευτικές πτήσεις ή μετάβαση προσωπικού σε ανθρωπιστικές αποστολές. Αυτές όλες οι πτήσεις εξαιρούνται από το πρόγραμμα ε, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Ε, σε γενικές λοιπόν γραμμές ε, υπάρχουν δύο-τρία βασικά θέματα και επιβεβαιώνουμε ότι κατά την άποψή μας μπορούμε να εισάγουμε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς στηρίζουμε την Επίτροπο και την ομάδα που ήταν στο Μουντράλ, στον ΙΚΑΟ, αλλά και τα κράτη-μέλη. Είμαστε ιδιαίτεροι αισιόδοξοι, γιατί ο πρωταρχικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι να ανασταλεί η απόφαση. Ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά τους ε, σκιώδης ηγητές για τις πολύ συζητήσεις και ευχαριστώ και όσους από την Επιτροπή πρότειναν το σχέδιο αυτό. Ε, Περιμένω περιμένω τα σχόλιά Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Βίμ Κάμπ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ εδώ τον Μάρκος Βέρμπερ, ο οποίος ε, ε, δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Εξ του λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Φώστερε, ε, για την εξαιρετικά επικοδομητική της ε, εργασία, ε, εργασία την οποία έφερε εις πέρα στους τελευταίους μήνες. Πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες αυτής της πρότασης παρουσιάστηκαν πάρα πολύ σωστά από την κυρία Φώστερ τα προηγούμενα πέντε λεπτά ε, εμείς έχουμε υποβάλει κάποιες συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες ε, και, και νομίζω ότι μπορεί να τις υποστηρίξει. Ε, συμφωνώ με την κυρία Φώστερ όταν λέει ότι επί του θέματος αυτού θα πρέπει να αποφύγουμε να πάρουμε πολύ διαφορετικές και μοιρασμένες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν μελετήσουμε τα όσα έλαβαν χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάναμε ε, πολλά όσον αφορά την ανταλλαγή εκπομπών. Θα πρέπει να προχωρήσει η πρόοδος όμως ε, η Επιτροπή ΕΝΒΗ ελπίζω ότι προσεκτικά θα μελετήσει την γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών που είναι πολύ ε, σοφή και ε, σόφρον και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και θέση του συνόλου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ο επόμενος ομιλητής Ευχαριστώ πολύ. Όταν είμαστε στο Μόντρεαλ το προηγούμενο ε, φθινόπορο ε, δουλέψαμε ε, σε καλή συνεργασία και μιλήσαμε και για τα κατόφλια και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα είναι σαφή και νομίζω ότι οφείλουμε να διαπιστώσουμε το εξή ότι θα πρέπει στην Ευρώπη τώρα να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε ε, να έχουμε ένα συνολικό σύστημα το οποίο και θα θεσπιστεί και θα λειτουργεί σωστά. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε το σύστημα το οποίο εμείς ε, θα υλοποιήσουμε να συνδυάζεται καλά με το συνολικό, χωρίς τριβές και χωρίς ε, προβληματισμούς. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση είναι θετική έτσι όπως παρουσιάστηκε γιατί πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό είναι το σωστό γιατί η Ευρώπη πρέπει να προσπαθήσει να ε, κάνει, να καταστήσει πιο ε, ισχυρό το παγκόσμιο σύστημα. Εδώ μπορούμε να αποφασίσουμε τι είδο σύστημα θέλουμε και πρέπει να το κάνουμε με τρόπο ώστε να ενισχύσουμε το συνολικό σύστημα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και η απαραίτητη πολιτική βούληση έτσι ώστε να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία έχουν καθοριστεί από τη Συμφωνία των Παρισίων δεν είναι δυνατόν ε, να ε, ξεχάσουμε αυτό το ζήτημα της αεροπλοείας ε, όταν μιλάμε για το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλη, ολόκληρη την πρόταση, αλλά συμφωνούμε με τα περισσότερα σημεία. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και προτάσεις από τους πράσινους και την ΚΟΕ που εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστές και θα πρέπει να στηριχτούν. Ε, είναι κρίμα που οι προτάσεις ε, της ΓΚΟΕ έμειναν έξω από σχεδόν όλες ε, τις συμβιβαστικές προτάσεις. Νομίζω ότι το, το ζήτημα της Τις δημοπρασίες και τα χρήματα από τις δημοπρασίες ε, των εκπομπών θα πρέπει να χρηματοδοτούν όχι γενικά την έρευνα αλλά την έρευνα για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή. Ε, κατά τα ε, λοιπά αναλύουμε τον κατάλογο ψηφοφορίας και θα ψηφίσουμε αναλόγως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας, να ευχαριστώ θερμά την κυρία Φώστερ. Εργαστήκαμε πάρα πολύ καλά, αναφέρθηκε ήδη ότι υπάρχουν οκτώ συμβαστικές προτάσεις. Οι φιλελεύθεροι στηρίζουν όλες αυτές τις ε, προτάσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς ασχολούμαστε εδώ και πολύ καιρό με αυτό το σύστημα της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής. Η δική μας η πολιτική ομάδα, όπως είπε πολύ σωστά, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια λύση, γιατί έτσι κι αλλιώς ε, έχουμε παγκόσμια οι μεταφορές, σε διεθνές βεληνικέ. Ο ΙΚΑΟ, ίσως εκεί μπορούμε να ασκήσουμε λιγάκι πίεση στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, να προσπαθήσει ο ΙΚΑΟ να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει αποφασίσει. Συμμετέχουν όλοι, ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το θέμα είναι κατά πόσον θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Και θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα, όσο και να το θέλαμε, να θέσουμε περισσότερο φιλόδοξο φιλόδοξα σχέδια ως Ευρωπαίοι. Γιατί αν το κάνουμε είναι δυσάρεστο μετά οι άλλοι να αρνηθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι σε διεθνή κλίμακα να συμβαδίσουμε με τον ΙΚΑΟ, να σκίσουμε πίεση και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω το είναι και οι πράσινοι να συμπεριληφθούν και άλλες εκπομπές, όχι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα. Ε, Βεβαίω το διοξείδιο του άνθρακα είναι το σημαντικότερο και ίσως θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποιο άλλο, κάποια άλλη οδό. Οι φιλελεύθεροι στηρίζουν τις τροπολογίες και την έκθεση και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοδομητική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ε, η κυρία Κίλενεν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο κυρία Φώστερ για την ε, πολύ επικοδομητική συνεργασία. Πρέπει να πω ότι ίσως ε, η φιλοδοξία μας ε, ή το επίπεδο φιλοδοξίας που έχουμε διαφέρει. Ωστόσο, ε, νομίζω ότι η στάση μας είναι σαφής μέσω των ε, τροπολογιών. Ωστόσο, το σημείο κίνησης είναι κοινό. Τη Συμφωνία των Παρισίων μας υποχρεώνει ε, να δράσουμε. Και ήλπιζα ότι στις θαλάσσιες ε, μεταφορές ε, ε, θα είχαμε τουλάχιστον, μάλλον στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, θα είχαμε μια καλή συμφωνία όπως και στις θαλάσσιες μεταφορές. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση όπως έγινε άλλωστε και στον τομέα των μεταφορών, των θελασσίων μεταφορών. Παραμένει βεβαίως ε, ένα μεγάλο ερώτημα στην δική μας ε, οικογένεια, ε, δηλαδή η ανάπτυξη του ενιαίου ουρανού, γιατί προχωράει με εξαιρετικά αργό ρυθμό και πρέπει πρώτα να δούμε τα οίκο μας πριν αρχίσουμε να καθαρίζουμε ή να προσπαθούμε να λύσουμε τα παραπέρα θα πρέπει να δούμε εάν μπορούμε να βρούμε και ε, λύσεις σε τοπικό επίπεδο ε, πριν ε, συνδράμουμε μέσω κοινών λύσεων. Εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές πιστεύουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί το κείμενο και ελπίζουμε ότι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα, μας, θα λάβουν υπόψη την Εν πάση περιπτώσει είναι γεγονό ότι εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλες τις συμβιβαστικές λύσεις γιατί μερικές φορές είναι εξαιρετικά αδύναμα αυτά τα ε, συμβιβαστικά κείμενα. Ωστόσο θα ευχαριστήσω την κυρία Φώστερ ε, γιατί επιδιώκουμε όλοι ένα κοινό στόχο και η συνεργασία ήταν πολύ καλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank Σας ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, μιλάμε εδώ και συνεχώς αυξάνονται οι εκπομπές στον τομέα της αεροπλοείας. Και τώρα αποφασίσαμε να στείλουμε τις αποφάσεις ε, για να μειωθούν οι εκπομπές. Όμως κατά την άποψή μας ε, οι αποφάσεις θα έπρεπε να έχουν ληφθεί εχθές. Και όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων το 2021, το 50% θα έπρεπε να είναι το ανώτατο όριο όσον αφορά τις πτήσεις από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να διευκολύνουμε και την εφαρμογή του προγράμματος που έχει αποφασίσει ο ΙΚΑΟ. Ε, κάτι άλλο, ο ΙΚΑΟ έχει καθορίσει κάποια όρια, ε, δεν είναι τα καλύτερα, αλλά καλύτερα από το τίποτα. Όσοι λοιπόν συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τα ανώτατα όρια. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτά τα κεντρικά, όπως αναφέρονται μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται μέσα από το σύστημα της κατηγορίες δικαιωμάτων εκπομπή. Οι ενδοενωσιακέ πτήσει θα πρέπει να είναι κάτω από το όριο, το ανώτατο όριο τη εμπορία δικαιωμάτων εκπομπή. Εξάλλου η αεροπλοεία έχει πολλέ επιπτώσει το θείο, ε, οξύδια του θείου και πολλά άλλα εκλείονται, αλλά ο ΙΚΑΟ ορίζει ότι η εκπομπές από την, στην αεροπλοεία είναι υπόλοιπε, πολύ μεγαλύτερες, διπλάσιες τουλάχιστον από ότι αυτές του διοξιδίου του άνθρακα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ισχύει ένας πολλαπλασιαστής όσον αφορά τις εκπομπές από την αεροπλοεία. Θα πρέπει να ισχύει εξάλλου και η αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Εμείς θεωρούμε ότι αν δεν υπάρχουν ανώτατα όρια αυτό δεν θα οδηγήσει στο να μειωθούν εκπομπές και επίσης ε, θα καταστεί δυνατό να χαθούν αρκετά χρήματα. Η αεροπλοεία δεν αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα ε, διαρροής του άνθρακα όπως ε, σε άλλους τομείς. Ως εκ τούτου θα πρέπει όλες οι εκπομπές να είναι αντικείμενο δημοπρασίας. Εμείς συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει όμως ένας γραμμικός παράγων από το 2021 και πιστεύουμε και ότι όλα τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, στρέφομαι πλέον προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λοράνς Γκράφ. Ακούσατε τις απόψεις ε, είχαμε πολλές συζητήσεις ε, επί της ε, κλιματικής συμφωνίας, είχαμε και τα τελευταία νέα από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και είναι σαφές το ότι οι συνάδελφοι είναι πιο απαιτητικοί, έχουν απαιτήσει, επίσης κρούν το κόδωνα του κινδύνου, πρέπει η Ευρώπη να καλύψει κενά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ναι, όντως ακούσαμε προσεκτικά τις απόψεις θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την κυρία Φώστερ, την εισηγήτρια, αλλά και τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, είναι καλό που ακούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχατε καλές ε, ε, συζητήσεις. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει γρήγορα να προχωρήσουμε στον φάκελο αυτό. Επομένως, Περιμένουμε ε, με μεγάλη αδημονία τις ε, προτάσεις σας και τις συμβαστικές σας ε, προτάσεις έτσι ώστε να μπορέσει να εγκριθεί η πρόταση μέχρι το τέλος του έτους γιατί αυτό είναι απαραίτητο όσον αφορά την επέκταση του, του, του πρόσκαιρου πεδίου εφαρμογής τα τρία χρόνια ναι όντως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για το συνολικό σχέδιο έτσι ώστε να μπορέσει δηλαδή να γίνει έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ε, ε, επιχειρησιακά ε, έτοιμο. Κατά αυτή την έννοια, ήδη πολλή δουλειά γίνεται στα πλαίσια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και επίσης Επίσης ε, ζητούμε και περισσότερες πληροφορίες ε, σχετικά με το κατά πόσον και με ποιο τρόπο χώρες οι οποίες έχουν ήδη δεσμευτεί ε, με το πρώτο επίπεδο θα προχωρήσουν στην εφαρμογή και του δευτέρου επίπεδου. Βεβαίω ε, ε, πρέπει να ακούσουμε, να περιμένουμε και τα νέα από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, μέχρι τώρα αυτά που μας κοινοποιούνται δεν πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται, περιμένουμε και να δούμε και ποια θα είναι, ποιες θα είναι και οι προθέσεις τη Κίνα. Ωστόσο, α μην προδικάζουμε. Θα περιμένουμε να δούμε έτσι ώστε να έχουμε μια σαφή ε, εικόνα και για το πρόγραμμα Κορσία και το πώς θα ε, υλοποιηθεί. Ε, με την ίδια προσοχή θα πρέπει να δούμε και τις ε, εσωτερικές εντός ε, Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πτήσεις και τις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις υπό την Συμφωνία των Παρισίων και γνωρίζετε ότι βεβαίως όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην προκειμένη περίπτωση των εκπομπών της αεροπορίας και τουλάχιστον να έχουμε να φτάσουμε στο 40% που αφορά την εγχώρια μείωση των ε, ε, εκπομπών. Από τη μία μεριά βέβαια ε, έχουμε και στα πλαίσια του Κορσία την ε, προσπάθεια η οποία γίνεται όσον αφορά τη μείωση ε, σε εγχώριο επίπεδο των εκπομπών. Από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε και τις διεθνείς ε, συμφωνίες και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα στοιχεία αυτά. Η συγκυρία είναι τέτοια που οι συμφωνίες των Παρισίων και μετά από τις δηλώσεις Τραμπ αποκτούν πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης να πω ότι την αναφορά στον, ε, ε, στον παράγοντα γραμμικής ε, μείωσης μπορούμε να τον εντάξουμε στο κείμενο, πάντως θα περιμένουμε να λάβουμε τα συμβιβαστικά σας κείμενα, τις συμβιβαστικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω τώρα το λόγο στην κυρία Φώστερ. Um, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι αυτά που ελέγχθησαν από το και ήταν πολύ σωστά να τεθεί το θέμα έγκαιρα, διότι τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια ο τομέας της αεροπλοείας έχει συμβάλει τα μάλα στις ε, εκπομπές. Εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, ήμουν και εισηγήτρια για τον νέο ευρωπαϊκό ουρανό. Ξέρω πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν ε, και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αμβλύνουμε τις εκπομπές. Εξάλλου, Μιλάμε για περίπου 4 δις που χρησιμοποιήθηκαν για τον ενιαίο ευρωπαϊκό όρο. 1,4 δις μάλλον. Ε, υπάρχει μια συμφωνία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό όρανο. Άρα γίνονται πάρα πολλά. Τώρα πλέον αναπόκειται στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τις ε, δυνατότητές τους γιατί διαμαρτύρονται αλλά πρέπει μόνα τους να φροντίσουν ε, έτσι ώστε να μην στέλνουν τα αεροσκάφη να περιμένουν παραδείγματο χάνει δύο ώρε στο αεροδρόμιο του Λονδίνου. αυτά που είπε ο συνάδελφο από τον Ελισάν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο ότι ξέρουμε ποια είναι η συμφωνία του Παρισιού. Ε, θεωρώ ότι επ' αυτού Υπάρχουν κάποιες ε, ε, παλινδρομήσεις, αναφέρετε τις ΗΠΑ και είπατε ότι προφανώς οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία. Όμως εγώ να σας πω κάτι θετικό. Επειδή δεν εντάσσεται η αεροπλοεία και οι θελές μεταφορές στη Συμφωνία του Παρισιού, εκεί θα μπορούσαν τουλάχιστον να προσχωρήσουν οι ΗΠΑ γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι η Συμφωνία του Παρισιού. Αυτό λοιπόν είναι ένα καλό σημείο διαπραγματεύσεων, αν συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την έρευνα, όταν μιλάμε για την κατοχήρωση πόρων για αυτά τα προγράμματα. Πρόκειται για προγράμματα που βασίζονται στην έρευνα και σας είπα ότι θα πρέπει να συμμετέχει η βιομηχανία αν θέλουμε να αμβλύνουμε τις ε, εκπομπές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα σχόλια από τους φιλελεύθερους, να ευχαριστήσω την κυρία Κιλίνεν, την φίλη και συνάδελφο. Δυστυχώς ε, αναφέρθηκε και από, τη, από τον συνάδελφο από τους Πράσινους, πράγματι ε, είπανε ας έχουμε μια ευρωπαϊκή λύση. Είχαμε ευρωπαϊκή λύση και εδώ και δέκα χρόνια βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζεται αυτή η ευρωπαϊκή λύση. Άρα η καλύτερη λύση είναι να επιτύχουμε λύση σε παγκόσμιο βελινεκές. Αυτή είναι η δική μου η πρόταση και αναφέρομαι πάλι στο συνάδελφο από του πράσινου. Μα δεν μπορείτε να περιμένετε τα κράτη-μέλη και οι εταιρείε να λειτουργούν διαφορετικά συστήματα για εσωτερικέ πτήσει, για πτήσει σε τρίτε χώρε. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα, να δώσουμε στους αρμόδιους τα εργαλεία να κάνουν δουλειά τους και ας προχωρήσουμε. Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα που ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή επικοδομητική λύση και πράγματι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φώστερ. Αύριο το πρωί θα γίνει η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Συνεχίζουμε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την πρόταση της Κομισιόν για την αναδιατύπωση της οδηγίας του 2009 όσον αφορά την πρόθεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή η πρόταση συνδέεται με τις προτάσεις αναδιατύπωσης του τρίτου ενεργειακού πακέτου, καθώς επίσης και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, ε, βάσει των συμφωνιών των Παρισίων 2015. Ένα από τα κεντρικά στοιχεία κλειδιά βεβαίως είναι η διαφοροποίηση του τομέα των μεταφορών και η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Σε αυτού του σημείου η Επιτροπή μας θα δώσει τη γνωμοδότησή της στην Επιτροπή Ήτρε και θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Αϊκχούτ για να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση του κυρία Αϊκχούτ. Κύριε εισηγητά, έχετε την, ε, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε. Πράγματι πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά θέματα του πακέτου που κοινοποίησε πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέματα ε, κλίματος, με θέματα αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και βέβαια αναδιατύπωση της νομοθεσίας για την ανάπτυξη των ανανεωσίμων ενεργειών από το 2021 έως το 2030. Χρειαζόμαστε όλο αυτό το φάσμα των ανανεωσίμων ενεργειών και στον τομέα των μεταφορών που παίζει σημαντικό ρόλο διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το 32% της ενέργειας και, από, και κλείουν στην ατμόσφαιρα 22% των συνολικών αερίων θερμοκηπίου. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Πολλές από τις συζητήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στρέφονται γύρω από τους στόχους για τις ανανεώσιμες ενέργειες συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 24% μέχρι το 2030. Υπάρχει κοινή κατανόηση όμως εδώ στο Κοινοβούλιο ότι ο πύχης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και για, για να φτάσουμε στο 20% το 2020 θα πρέπει να έχουμε ετήσια αύξηση 5% της χρήσης ανανεωσίμων μέχρι το 2020 και μετά από το 2020 για να φτάσουμε στο 27% μέχρι το 2030 θέλουμε 1% ετησίως αύξηση χρήσης ανανεωσίμων. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι όταν οι ανανεώσιμες γίνονται πλέον ανταγωνιστικές και αν εξετάσετε τις διάφορες τιμές των ε, ενεργειακών πόρων θα δείτε η Κομισιόν να προτείνει να κατέβει από την ετήσια αύξηση από το 5% στο 1% μετά το 2030. Δεν νομίζω να το βλέπουν πολύ ανθρωπιλογικό αυτό το πράγμα. Μέσα στο Κοινοβούλιο θα συζητηθεί πολύ το ενδεχόμενο αύξηση του στόχου αυτού. Το βάζω και στην εκθεσή μου. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι πρόκειται κυρίως για αρμοδιότητα της Επιτροπής Ενέργειας, αλλά επειδή τέλο πάντων όλες οι επιτροπές προβάλλουν τα δικά τους και άλλη μια συζήτηση που υπερβαίνει τα όρια της παρούσας Επιτροπής είναι αν θα χρειαστούμε εθνικούς στόχους, ναι ή όχι. Γνωρίζουμε ότι εντός του Συμβουλίου αναπτύχθηκε μια συμφωνία κυρίων για να διευκολυνθεί ιδίω οι Βρετανοί, οι οποίοι δεν θέλαν να ακούσουν περί ανανεωσίμων, και για να φτάσουν σε κάποιο συμβασμό βάλαμε ευρωπαϊκό στόχο για τι ανανεώσιμε, αλλά όχι εθνικού στόχου. Αυτό είναι μια από εκείνε τι περίφημε συμβαστικέ ευρωπαϊκέ λύσει μεταξύ χωρών μελών. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο σωστό δρόμο να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ο συμβασμό αυτό προκαλεί έτσι πλέον ασάφεια και μετά προχωρεί η συζήτηση για θέματα διακυβέρνηση Είναι πολύ καλύτερο να υπάρχουν εθνικοί στοχοί και η ιστορία έχει δείξει άλλωστε ότι οι εθνικοί στόχοι παρακινούν τι χώρε, όπω βλέπετε την Ολλανδία, όπου δεν θα είχε υπάρξει προτριετία συμφωνία για την ενέργεια εάν δεν υπήρχαν εθνικοί στόχοι επιβλημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να παραταθούν και να συνεχιστούν οι εθνικοί στόχοι. Είναι λογικό αυτό. Και αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε αργότερα και με το Συμβούλιο. Αυτά είναι με λίγα λόγια οι συζητήσει που θα χρειαστεί να κάνουμε για τη νέα οδηγία περί ανανοσίμων. Υπάρχει και ένα μέγα μέρος ειδικότερα για τις μεταφορές. Εκεί θα χρειαστεί να κινηθούμε σύντομα στη συζήτηση περί βιολογικών καυσίμων. Πρώτα όμως, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λίγο πολύ για την πρώτη γενιά βιολογικών καυσίμων. Υπάρχει ήδη ένα νότατο όριο 7% πρόκειται για ε, σταδιακή μείωση μέχρι το 3,8% το 2030. Είμαι βέβαιος ότι θα χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ αποφάσισα να μην αλλάξω τον στόχο αυτό. Διατηρώ το 3,8% στην γνωμοδότησή μου. Γνωρίζω ότι άλλοι επιθυμούν να δουν πλήρη σταδιακή κατάργηση. Θα έχουμε λοιπόν επιτάπητος όλες τις ενδεχόμενες επιλογές. Ο λόγος για τον οποίο εμένω και εγώ στο 3,8% είναι ότι είναι ισχυρή επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν προκειμένου. Αυτό που δεν μου αρέσει με τον στόχο αυτό είναι ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση ε, μαύρου-άσπρου, δηλαδή χωρίς ενδιάμεσες αποχρώσεις για, τις, ε, για τα βιολογικά κάψιμα που έρχονται από καλλιέργειες. Και δεν είναι απαραίτητα κακά όλα αυτά προτιμά και ο εισηγητής να υπάρχουν σαφή ισχυρά κριτήρια επιτάπητος και αυτά, στη βάση αυτά, αυτών μπορούμε να δούμε ποια πράγματα έχουν καλά τα βιολογικά κάψιμα και ποια όχι. Θα υπάρξει μια αρνητική επίπτωση στο βιολογικό δίζελ. το γνωρίζω αυτό, αλλά τα βιολογικά καύσιμα που προέρχονται από καλλιέργειες, στο βιολογικό δίζελ, δεν τα πάνε πολύ καλά και έχουν συχνά και αρνητική επίπτωση στα αέρια θερμοκηπίου. Ένα παράδειγμα είναι το λάδι από το φινικέλαιο. Είναι το φινικέλαιο. Ε, ε, γνωρίζω ότι οι ορισμένοι ζητούν να καταργηθεί πλήρως το φινικέλαιο ως η χρήση του δηλαδή στο βιολογικό καύσιμο. Είναι δύσκολο να πει κανείς για ένα μόνο πράγμα δεν το θέλουμε καθόλου. Εγώ προτιμώ όπως είπα να υπάρξουν ξεκάθαρα κριτήρια και τότε θα δείτε ότι τα ανεπαρκή ή τα κατάλληλα καύσιμα θα βγουν από μόνα τους λόγω των κριτηρίων από το σύστημα. Το φινικέλαιο δεν θα μπορέσει να παραμείνει μέσα στις βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές. Ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί χώρο για τα καλά βιολογικά καύσιμα να μπορούν να πιάσουν περισσότερο χώρο μέσα σε αυτό το στόχο 3,8% διότι λέει η Κομισιόν ότι το 3,8% καταστρέφει λίγο πολύ τις καλλιέργειες βιολογικών καυσίμων. Θα δείτε ότι ορισμένα από τα κακά καύσιμα αυτά θα εκπέσουν. Βλέπω ότι βιάζεται η Πρόεδρος. Θα μπορούσα να σας μιλώ για μια ώρα, αλλά θα επιταχύνω, σύμφωνοι. Με τις προτάσεις αυτές πετάμε έξω τα κακά βιολογικά καύσιμα και αφήνουμε χώρο κάτω από το ΚΑΠ, κάτω από το το όριο του 3,8% για τις εθανόλες, που είναι για την ώρα στο 20% του συνόλου των βιολογικών καυσίμων ε, πρώτης γενεάς. Και μετά προχωρούμε στα προηγμένα βιολογικά καύσιμα, που έχουμε τα προηγμένα, έχουμε ε, ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμα, ανανεώσιμες ενέργειες και αυτά θα πρέπει να φτάσουν στο 6,8%. Έχουμε λοιπόν ένα πρώτο όριο 3,8% και μετά ένα 6,8%. Ο εισηγητής αφαιρεί την πρόταση της Κομισιόν ώστε να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός όλων των υπολείπων καυσίμων που θα κινηθούν μέχρι το όριο του 6,8%. Ο δε εισηγητής κάνει και ορισμένε προτάσει για να διασφαλίσει ώστε ο ανταγωνισμό μεταξύ τη ε, ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμα και τα βιολογικά να είναι κάπω ισορροπημένα. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα που προέρχονται από απορρίμματα, ναι. Ε, και αυτό το θέμα ε, θα ε, αντικαταστήσουν σιγά σιγά τα ορυκτά καύσιμα. Προχωρεί γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν τέλει να υποβάλει μια καλύτερα διατυπωμένη πρόταση για τα ορυκτά καύσιμα που παράγονται από απόβλητα. Εν τέλει, η ερώτηση είναι ποια είναι τα προηγμένα βιολογικά καύσιμα που όλοι θέλουν να ε, τα παράγουν. Όλοι θέλουν να έχουν βελτιωμένα ε, ε, προηγμένα βιολογικά καύσιμα. Υπάρχουν εφαρμογές αυτών και εκτός ενέργειας και εκτός μεταφορών. Άκουσα βιομηχανικούς φορείς που ήρθαν στο γραφείο μου να με δουν να μου λένε ότι οι επιδοτήσεις που θεωρούν τώρα, θεωρούνται ότι πηγαίνουν για προηγμένα βιολογικά καύσιμα χρησιμοποιούνται από τη χημική βιομηχανία για άλλες χρήσεις. Και αυτό που βλέπουν είναι ότι λόγω αυτής της προώθησης προς τα βιολογικά καύσιμα κινούνται προς τα βιολογικά καύσιμα και αυτοί ως βιομηχανικοί φορείς αναγκάζονται εν τέλει να χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα. Για παράδειγμα φινικέλαιο. Να το που ξεπηδά πάλι το φινικέλαιο. Επομένω τίποτε δεν είναι δωρεάν. Θα χρειαστεί να δούμε και τα προηγουμένα βιολογικά καύσιμα για να μην επαναλάβουμε το ίδιο λάθος που κάναμε με τα καύσιμα, με βιολογικά καύσιμα πρώτης γενεάς και εκεί πρέπει να ισχύσουν λοιπόν ε, κριτήρια βιωσιμότητα. Εν τέλει, αεροπορικέ μεταφορέ. Χρησιμοποιεί κάποιου πολλαπλασιαστέ που δεν βρίσκονται ότι είναι σωστή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν υπάρχει ένα τομέα όπου τα βιολογικά καύσιμα και τα προηγουμένα βιολογικά καύσιμα θα πρέπει πράγματι να αναπτυχθούν, είναι ασφαλώ η αεροπλοεία. Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν εκεί εναλλακτικά καύσιμα. Γι' αυτό ο εισηγητή προτείνει να μπει η αεροπλοεία καθαρά, ρητά, μέσα στο στόχο του 6,8%. ώστε τις μεταφορές όπου υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει τώρα ε, πιο δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ προηγουμένων βιολογικών καυσίμων και ανανεώσιμου ηλεκτρικού ρεύματος, να μπει και η ε, αεροπορική, ε, το μέσο αεροπορικών μεταφορών. Αυτή είναι η λογική που ακολουθεί η πρόταση που αλλάζει λίγο, η δική μου δηλαδή, που αλλάζει λίγο την πρόταση τη ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω ότι είναι θετική και αναμένω τις αντιδράσει. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Ατσεκούτ. Ε, είναι πραγματικά μεταδοτικό το πάθος σας και με πάθος σας ακούμε, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας. Δίνω το λόγο στους Σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε στην αρχική φάση της συζήτησης. Ε, πρέπει να πω ότι ε, έχω κάποιες, κάποιους προβληματισμούς ε, παρόμοιους ε, με του ε, συναδέλφου και όσον αφορά την πρόταση και όσον αφορά ε, συγκεκριμένες, συγκεκριμένα μέτρα ή είδη μεταφορών. Πολλές λέω από, αυτά, από αυτούς τους προβληματισμούς τους έχω και εγώ ταυτόσιμους. Όσον αφορά τώρα το ποσοστό το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτικό για τις μεμονωμένες χώρες αλλά θα είναι ευρωπαϊκός στόχος, εδώ ε, εδώ θα πρέπει να υποβάλουμε το σύνηθες ερώτημα, δηλαδή ποιες είναι οι χώρες οι οποίες ε, θα εφαρμόσουν και ποιες είναι οι χώρες οι οποίες ε, τελικά θα μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτήν την απέτηση. Σωστή, σωστό λοιπόν το ερώτημα και όχι μόνο, και δεν ισχύει μόνο για τον τομέα των μεταφορών, θα πρέπει να το δουλέψουμε, να το μελετήσουμε αυτό. Ε, τώρα, στα πλαίσια του μείγματος ε, δεν ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε με την αύξηση του στόχου μέχρι το 40% έτσι ώστε να γίνει βιώσιμο όλο το ζήτημα. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι για να είναι βιώσιμος ένας στόχος θα πρέπει να είναι βιώσιμος και σε διάρκεια χρόνου και όχι και σε βάθος χρόνου και όχι μονάχα λόγω του μίξε αλλά και γιατί δίνεται η δυνατότητα από όλους τους τομείς ε, να προωθηθεί η αηφορία αυτού του στόχου. Νομίζω ότι οπωσδήποτε πέρα από τα όσα ωραία μπορεί να πούμε θα πρέπει να είμαστε και αρελιστές. Όσον αφορά το τομέα των μεταφορών, ε, ο στόχος του 10% που είχε ε, πρωτήτερα αναφερθεί και που δεν υπάρχει πλέον μετά το 2020, η συζήτηση είναι ανοιχτή πάνω σε αυτό. δεν είναι σίγουρο ότι είναι σίγουρα καλός στόχος να αφαιρεθεί αυτό το 10% από τις μεταφορές. Ε, θα δούμε τώρα ποιες θα είναι οι μελλοντικές προτάσεις οι οποίες θα προκύψουν. Επίσης, ορθώς υπογραμμίζεται, την αστεριζόμαστε και εμείς σαν Επιτροπή Μεταφορών, ε, όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, ο εισηγητής ε, μελέτησε ενδελεχώς τους διάφορους υποστόχους. Δεν θα επιστρέψω σε αυτό, αλλά συμμερίζομαι και εγώ το ερώτημα του εισηγητού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν προτείνει το πέρασμα από τα βιοκαύσιμα πρώτη σε βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Είναι απόλυτα ανοιχτό το θέμα, ε, προέρχεται από, πολλές, από πολλούς κλάδους, διατροφική βιομηχανία, ε, χημική βιομηχανία και τα λοιπά και σε σχέση ειδικά με το ε, παράρτημα, το διαβόητο παράρτημα 9 πρέπει να πω ότι χρησιμοποιείται ήδη ε, και στον τομέα των τροφίμων και στο τομέα της παραγωγής ε, ε, ε, ζωοτροφών και στον χημικό τομέα, όπως έλεγα και προηγουμένως, ε, η χρήση ας πούμε για παραγωγή βιοκαυσίμων, χρήση για παραγωγή βιοκαυσίμων θα μπορούσε να προκαλέσει και ανισορροπίες αλλά και οπωσδήποτε μάχη όσον αφορά τις τιμές. Τώρα όσον αφορά την ποσότητα του προϊόντος που θα πρέπει ε, να αφορά τα προηγμένα βιοκαύσιμα και αν και κατά πόσο μπορεί να καλύψει το σύνολο του, της ε, ζήτησης. Αυτό είναι ένα άλλο ε, ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε και τρόπους έτσι ώστε το έλλειμμα να αντισταθμιστεί. Αυτές είναι λίγες μόνο από τις ορισμένα μόνο από τα προβλήματα τα οποία μπορούν να συνδέονται συνδέονται με την ε, μείωση της χρήσης των λιπτών καυσίμων. Αυτά είναι τα κεντρικά θέματα και βεβαίως και η διασύνδεση με το φάκελο για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και το πέρασμα ε, σε προηγμένα βιοκαύσιμα τα λεγόμενα δεύτερης γενιάς. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν η υπόψη και θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη μας και τα αιτήματα των διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας. Ε, αυτά. Merci, euh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαβίνη. Θα ήθελα να σας ζητήσω να, είμαστε, ε, να είναι οι επόμενοι ομιλητές ε, πιο σύντομοι, γιατί περιμένουμε και την Επίτροπο Μεταφορών σε λίγο. Merci, ε, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή όσον αφορά τις ε, πρώτες προτάσεις ε, τροπολογιών του με τις οποίες συμφωνούμε. Στην ουσία ε, έχουμε εδώ ένα κείμενο το οποίο είναι ουσιώδου σημασία και που έχει πολύ συγκεκριμένο αντίκτυπο. Ας πούμε στο παράδειγμα του Ile de France σήμερα και αύριο έχουμε πολύ υψηλές εκπομπές οι οποίες συνδυαζόμενες με τις υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν ε, μεγάλα προβλήματα. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ευάλωτοι και μικρά παιδιά πρέπει να μείνουν ε, σε περιορισμό κατοίκων και επομένως ε, καταλαβαίνουμε ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πέρσι ψηφίσαμε τη συμφωνία του, του Παρισιού και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα δεν θα έρθουν σε μερικά χρόνια αλλά ήδη σήμερα τα βλέπουμε και τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να μην ε, ε, δημιουργηθούν ε, συνθήκες αντίστροφες ή που θα έχουν τα αντίθετα από τα ευκταία αποτελέσματα. Αυτό είναι σίγουρο. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να βρούμε, και αυτό είναι το, πιο σημαντικό στοιχείο, να βρούμε ένα μείγμα το οποίο να είναι σωστό. Και θα πρέπει βεβαίως να δούμε το θέμα πιο σφαιρικά και με τους συναδέλφους του περιβάλλοντος ε, και του συναδέλφου της Γεωργίας και της Ήτρε ε, και τα λοιπά. Ε, αυτά και θα υποβάλουμε και τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σμάκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και τον κύριο Έκχαουτ, εισηγητή της νομοδότησης Και να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου. 94% του τομέα των μεταφορών χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο. Οι χώρες μέλη που δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν το στόχο του 10% μέχρι το 2020, εφού ο τομέας των μεταφορών εκλείσει την ατμόσφαιρα 22% των ε, αερίων θερμοκηπίου, ενώ οι ανανεώσιμες ενέργειες βεβαίως και αποτελούν ένα σημαντικό νέο στοιχείο για την πρόληψη της αναθέρμανσης του κλίματος και την αλλαγή στην χρήση ενέργειας. Βεβαίως διεξάγεται και έρευνα που ε, θα οδηγήσει και σε απασχόληση, θα οδηγήσει και σε ασφάλεια προμήθειας των... της ενέργειας. Ο Μπά ω μέλος των, Πρασίνων έχει βεβαίω τι δικέ του πολιτικές πεπιθήσει, τις οποίες σέβομαι απολύτω τις περιλαμβάνει και στο κείμενό του, αλλά ίσως ορισμένες φορές οι επιθέσεις τον οδηγούν κάπως πολύ μακριά. Γι' αυτό θα ήθελα και εγώ ε, να περιλαμβάνω ορισμένα πράγματα. Βεβαίω υπάρχουν στην του πολλά καλά πράγματα, βιολογικά καύσιμα, ανανεώσιμες, ανανεώσιμο ρεύμα, ας το πούμε έτσι. Είναι, είμαι καταρχήν θετικός, αλλά έχω ορισμένες παρατηρήσεις. Εγώ και η πολιτική μου ομάδα θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι το 2030 θα πρέπει να ισχύσει ο στόχος του 27% ανανεωσίμων ενεργειών στο σύνολο της χρήσης ενέργειας, όπως άλλωστε το έχει συζητήσει και το Συμβούλιο Ευρωών. Για μας είναι αναγκαίο να υπάρχει και μια ευκαμψία υπέρ των χωρών μελών και η αρμοδιότητα να αποφασίζουν για το δικό τους ενεργειακό μίξ. Η πρόταση να πάει ο στόχος στο 45% και μάλιστα να γίνει και δεσμευτικό στόχος για τις χώρες μέλη, ε, ε αυτό δεν μας βρέχει σύμφωνος. Επίσης, δεν είμαστε σύμφωνοι με την ιδέα οι υποχρώσεις για τα προηγμένα ε, βιολογικά καύσιμα να, περιστούν, να ξεπεράσουν μάλλον τον τομέα των μεταφορών. Για το τομέα των μεταφορών υπάρχουν ήδη ε, πολλοί περιορισμοί, επιβάλλονται ήδη πολλοί περιορισμοί και ίσω και υπερβολικά πολλοί περιορισμοί. Το λέω δέχεται αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όμως νομίζω ότι εδώ είναι λάθος να προσθέτουν και άλλοι περιορισμοί. Μετά θέλω να έρθω και σε αυτή την ε, ιδέα της διατήρησης της αξίας. Ε, ένας ένα ε, καύσιμο όπως η μελάσα που χρησιμοποιείται σε ορισμένου τομεί. Να μπει σε ανάμειξη με βιολογικά καύσιμα νομίζω δίνει λάθος μήνυμα. Έχουμε και άλλες παρατηρήσεις κύριε Πρόεδρε. Βέβαια θα τις διατυπώσω σε τροπολογίες. Πάντως ε, αναμένω επικοδομητική συνεργασία με τον κύριο Εκχάουτ. Ευχαριστώ κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ενεργειακή πολιτική είναι από τι πιο σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίνοντας από τις προτάσεις που έχουμε μπροστά μας, δεν βλέπω να έχουμε και μεγάλο λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Πολλά θέματα τέθηκαν σχετικά με την οδηγία και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών. Όπως είπε μόλις ο συνάδελφός μου, ο στόχος του 27% ανανεωσίμων ενεργειών μέχρι το 2030 δεν είναι αρκετά φιλόδοξος. Όμως, προωθεί και επενδύσεις της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων. Και θα προσελκύσει ακόμα περισσότερες επενδύσεις. Και το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη είναι σε θέση να τα επιτύχει αυτά είναι δυνατόν από την άλλη μεριά να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί εάν δεν είναι δεσμευτικοί για τις χώρες μέλη. Εδώ όμως ερχόμαστε σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας. Το ερώτημα είναι λοιπόν γιατί προσφέρει σε αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πολιτική θα πρέπει να είναι δυνατόν επιτευχθεί και να εφαρμοστεί και να δίνει και κάποιο στοιχείο ασφάλειας. Η ομάδα ALDE θα λάβει μια γενικότερη θέση γιατί τα θέματα είναι γενικά. Σε ό,τι αφορά τα ειδικότερα θέματα για, για την πολιτική μεταφορών, τίθεται το θέμα εάν οι στόχοι που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω είναι επιτεύξιμοι. και σε ό,τι αφορά τα ποσοστά των ε, καυσίμων δεύτερης γενναίας. Μπορούν να απαντηθούν οι ερωτήσεις αυτές. Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα θα αλλάζουν κάθε δύο χρόνια και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσθέτει διαρκώς νέες γενναίες βιολογικών καυσίμων. Διότι πόσο θα κοστίσει εν τέλει εάν εφαρμοστούν αυτά στις μεταφορές και άλλους τομείς. Πρέπει δηλαδή να δούμε και το κόστος των ιδεών αυτών που μόνες τους είναι καλές. Αλλά τέλος, η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές είναι λιγότερο αμφισβητούμενη από τη χρήση βιολογικών καυσίμων στις τροπολογίες που θα καταθέσω εξ ονόματος της ομάδας μου, των φιλελευθέρων δηλαδή, θα δώσω έμφαση στην χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, όπου αυτό είναι δυνατόν στις μεταφορές βέβαια. Ευχαριστώ. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτητα, γιατί πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Ε, και έχουμε συγκεκριμένη ώρα ε, για να έχουμε μια καλή ανταλλαγή απόψε με την ε, Επίτροπο η οποία είναι εδώ και η οποία ε, θα συμμετάσχει στην συζήτησή μας τώρα. Ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά που έκανες. Μπας. Θα ήθελα να πω ότι ε, θα πρέπει να δράσουμε με τρόπο ώστε όλοι οι τομείς της οικονομίας να συνεργαστούν υπό το πνεύμα της κυκλικής οικονομίας. Επομένως θα πρέπει να βρούμε και μία λύση να συμφωνήσουμε ε, σχετικά με το τι είναι πραγματικά απόβλητο, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή βιοκαυσίμων ή ε, αλλού. Επίσης, Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που κάνουμε βράχη πρόθεσμα έχουν μακροπρόθεσμα μεγάλη, μεγάλο αντίκτυπο ε, και στην ε, βιομηχανία και αλλού. Θα πρέπει να δούμε και τι ε, σχέση μπορεί να δημιουργηθεί με την πολιτική επιδοτήσεων και με την οικονομική πολιτική γενικότερα. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στον τομέα των καυσίμων. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κιλενέν. Θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Αγιόλα Σάντερ για ε, δύο λεπτά. Πολύ γρήγορα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάς για την έκθεσή του και κυρίως ε, γιατί γιατί κυρίως να υπάρχει μια ε, ισορροπία, γιατί διαφορετικά τα πράγματα ε, ε, είναι μια τρέλα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε ακόμα το κείμενο, θέλουμε επίσης να υπογραμμίσουμε ότι πραγματικά είναι επίγουσα η κατάσταση, να υπογραμμίσουμε επίσης ότι πολλές υποδομές δεν είναι έτοιμες και βεβαίως εμείς θέλουμε να υπάρξει ριζική αλλαγή και όσο γίνεται μεγαλύτερη εν πάση περιπτώσει η αλλαγή και όσο γίνεται πιο ε, νωρί. Επίσης στις αστικές ε, ζώνε χρειαζόμαστε ε, διαφοροποιημένη αντιμετώπιση γιατί υπάρχουν αστικές ζώνες για τις οποίε έχουν, ισχύουν κάποιοι άλλοι κανόνες ε, παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Επίσης ε, το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Συνδρομών μπορεί να ξαναδεί λίγο το θέμα έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να, αντιδράσουμε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ, είχα ζητήσει και εγώ το λόγο. σχετικά με τα καύσιμα, αγκοκαύσιμα, τη δεύτερη γενιά αυτών των καυσίμων, Πώς μπορούμε να έχουμε δεύτερη γενιά χωρίς να έχουμε την πρώτη. Αυτό θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Ε, όμως θέλω να πω και κάτι θετικό. Δηλαδή στη Γερμανία το 2000 αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να ισχύει ο νόμος ε, περί ανώσιμων πηγών ενέργειας. 4% ήταν τότε. Και οι πιο αισιόδοξοι είχαν σκεφτεί ότι αν φτάσουμε μετά από 15 χρόνια στο 10% θα ήταν πολύ καλά. Τώρα, μετά από 17 χρόνια, είμαστε στο 30% ε, με 4.000 νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ στην πυρηνική ενέργεια έχουμε 25.000 θέσεις απασχόλησης. Η κυβέρνηση λοιπόν τα πράγματα προχωράνε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να τα αναχαιτήσουμε, διότι ε, τα λιγνητορυχεία τα οποία εκπέμπουν περισσότερε εκπομπέ πρέπει να προστατευτούν. Θέλουν να προστατεύσουν τα λιγνητορυχεία για να μην υπάρχει τόσο μεγάλη και γρήγορη ανάπτυξη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχουν τεράστιε δυνατότητε. Αυτό αφορά την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι να θέλουν. Το είδαμε στη Γερμανία σε 17 χρόνια, από το 4% πήγαμε στο 30%, που είναι καταπληκτική επίδοση. Όλοι κερδίζουν από αυτήν και νομίζω όλοι θα πρέπει να προστατεύσουν προσανατολιστούμε προς τα εκεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα και να καλωσορίσω την κυρία Επίτροπο. Επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η πολιτική για τις εκπομπές είναι πολύ σύνθετη. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά να κάνουμε όσον αφορά την ε, μεταφορά των φορτηγών με συνδρομικέ μεταφορές. Ε, αυτό ακόμα δεν είναι ανταγωνιστικό. Υπάρχει και η δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές που θα κατατεθεί. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ε, θα δούμε τι κατεύθυνση θα καταδειχθεί. εγώ θέλω να στα, τοποθετηθώ στα βιοκαύσιμα και γενικότερα ε, στις ανώσιμες πηγές που ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, κερδοφόρηση φόρα. Ε, αυτό όμως ε, που χαρακτηρίζεται ως βιοκαύσιμο δεν ξέρω αν ήταν πάντα χρήσιμο για το περιβάλλον. Τροπολογία 25 όσον αφορά τη βιομάζα. Αναφέρεται από τον εισηγητή χρήσιμη βιομάζα, αλλά για να μεταφερθεί αυτά τα υλικά χρειάζονται ε, πολλές, ε, ένα, με, μεγάλες αποστάσεις οδικών μεταφορών, άρα δηλαδή και αυτές μολύνουν το περιβάλλον. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, κύριε Φίφερ. Σύντομα όμως, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με μεγάλη χαρά το ενδιαφέρον για αυτήν τη νέα οδηγία. Η αναθεώρηση της οδηγίας έχει ως στόχο ε, τα κρατημέλη μελη να ε, μπορέσουν να αναπτύξουν το δυναμικό τους και από κοινού να φτάσουν τουλάχιστον το 27% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Αυτό ε, περιλαμβάνει αρκετά μέτρα, όπως και τη δέσμευση η παροχή καυσίμων να τοποθετήσουν στην αγορά ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιοκαυσίμων, κυρίως βιοκαυσίμων. Επιτρέψτε μου κάποια σχόλια που αφορούν στο σχέδιο της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το στόχο. Ο στόχος που προτείνεται από την εισηγητή είναι συνεπής με το στόχο που είχε προταθεί στο σχέδιο της έκθεσης για τη διαχείριση, αλλά ε, μεγαλύτερος από το στόχο του κυρίου Μπλάνκο, εισηγητή της ε, Επιτροπής ε, Ήτρο και από αυτό που είχε προτείνει το Κοινοβούλιο σε παλαιότερα ψηφίσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θα παρακολουθήσει την όλη συζήτηση. Θέλει όμως να υπογραμμίσει ότι αν ε, υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια ε, αηφορίας, ίσως ε, είναι και δύσκολο να επιτευχθεί τελικά ο στόχος για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τα βιοκάψιμα. Η πρόταση περιλαμβάνει μια προσέγγιση που είναι να συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο αηφορίας ε, κριτήρια τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και αυτά ε, έχουν συζητηθεί παλαιότερα, παραδείγματος χάρη ε, στο πλαίσιο της οδηγίας ILOC. Η Κομισιόν ανησυχεί γιατί και οι έμεσες επιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Να τα κριτήρια της βιωσιμότητας ε, και της χρήσης γης ε, ίσως έχουν επιθύμητα αποτελέσματα κυρίως επειδή αυτά βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες που ακόμα όμως δεν είναι καταληκτικές. Επίσης, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η προτινόμενη έμεση, έμεσες επιπτώσεις ε, μπορούν να ε, παρεμποδίσουν στο μέλλον την χρήση βιοκαυσίμων που βασίζονται σε καλλιέργειες γιατί ενδεχομένως να μην επιτυχάνεται ο στόχος που είναι 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα αυτά πρέπει λοιπόν να τα σκεφτούμε πολύ προσεκτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα δώσω ένα λεπτό στον εισηγητή για να κάνει το συμπέρασμα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εγώ προσβλέπω στο να συνεργαστώ με όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Άκουσα ότι και αυτοί έχουν περίπου τις ίδιες ανησυχίες. Μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε. Ο Μάρκα ανέφερε θέμα της ε, μελάσας ε, στα βιοκαύσιμα για να είμαστε σίγουροι ότι ε, δεν θα χρησιμοποιείται για βιομηχανικές εφαρμογές. Και αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Κομισιόν ακόμα δεν έχει καταλήξει, αυτό το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον οποτεδήποτε αναφέρεται. Και τελικά ποιο αποφασίζει κατά πόσον τα πορίσματα της μελέτης είναι διαφεσβήτα ή όχι. Το μπορεί να ισχυριστεί κανείς και για την κλιματική αλλαγή. Με συγχωρείτε, η επιστήμη πάνω θα εξελίσσεται, θα προχωράει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Εγώ αυτό προτείνω και προσβλέπω στην ε, συζήτηση με τους σκιώδεις ηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει στις 27 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12. Περνάμε αμέσως ε, σε αυτό το οποίο αναμένεται όλοι, δηλαδή ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Μπελ την ε, ε, Επίτροπο. Καλώς ορίσατε κυρία Επίτροπε στην Επιτροπή μας. Κάθε φορά πρέπει να ομολογήσω που σας ζητούμε να έρθετε, είστε παρούσα. Ε, σήμερα θα στοχεύσουμε, θα εστιάσουμε μάλλον συγγνώμη τη συζήτησή μας ε, στο, στη δέσμη κινητικότητας ε, η οποία ε, υφίσταται έτσι εδώ και κάποιο διάστημα. Ξέρουμε ότι οι στόχοι είναι κοινοί, θέλουμε ε, και να καλύψουμε την εσωτερική αγορά, θέλουμε και τις, ε, ε, να καλύψουμε τους, τους όρους εργασίας των μισθωτών, θέλουμε να εντάξουμε και την ψηφιακή διάσταση, θέλουμε όλα και το περιβάλλον και επομένως θα σας δώσω το λόγο. Κυρία Επίτροπε, είμαι βεβαία ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες ε, οι συζητήσεις. 15 λεπτά λοιπόν θα έχετε. Στην αρχική σας εισήγηση και μετά θα έχουμε την μεθοδο ping pong συντονιστές σε 4 λεπτά. για να συζητήσουν με την Επίτροπο και μετά όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές, δύο λεπτά ο καθένας, θα ε, έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την ε, Επίτροπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πολύ προσοχή θα σας ακούσουμε. Και οι συντονιστές φαντάζομαι ότι είναι έτοιμοι να υποβάλουν πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Παρακαλώ κύριε Επίτροπο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτέ, αγαπητοί φίλοι, είναι πράγματι πολύ σημαντικό που βρίσκομαι σήμερα μεταξύ σας και μεγάλη τιμή, την οποία δράτω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία. την 31η Μαΐου έδωσε το πράσινο φως η Κομισιόν ε, για, το, για την ε, σημαντική αυτή δέσμη της κινητικότητας. Πριν όμως αναφερθώ σε λεπτομέρειες αυτής της δέσμης, θα ήθελα να μου δώσετε τη δυνατότητα να σας αναφέρω το ευρύτερο πλαίσιο ε, και να μοιραστώ μαζί σας κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά έτσι ώστε να κατανοήσετε το πλήρες εύρο, το πλήρες εύρος της εικόνας. Δύο στοιχεία λοιπόν δύο, όσον αφορά το πολιτικό ε, περιβάλλον ε, εξ αρχής η εντολή της ε, Κομισιόν ήταν ε, ε, δυνατή όσον αφορά την πιο δίκαιη και πιο ευρέα εσωτερική αγορά. Υπήρξαν θέματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά στην επίτευξη του στόχου αυτού της εμβάθυνσης της εσωτερικής αγοράς. τα σημεία που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση ε, και απόδοση της ε, ενέργειας, καθώς επίσης ε, και την δυνατότητα ανεξάρτητων πηγών ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ σημαντικά θέματα και από τη στιγμή που οι μεταφορές είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κατά κάποιο τρόπο διοξιδίου του άνθρακος και επομένως μόλυνσης έπρεπε οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ε, και ε, βεβαίως να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο του συνολικού στόχου της μείωσης των εκπομπών. Επίσης, η ψηφιακή αγορά και το ψηφιακό θεματολόγιο είναι πάντα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως τώρα οι διαθέσιμε τεχνολογίες είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο άρτιες και επομένως μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει χρησιμοποιήσει ψηφιακά ε, ε, εργαλεία έτσι ώστε να επιτύχει άλλους στόχους, έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και η εσωτερική αγορά αλλά και να αυξηθεί και η διασυνδεσιμότητα. Με τις δέσμες μας ε, ε, εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε τα θέματα. Το ίδιο κάναμε και με την δέσμη κινητικότητας. Ε, η προετοιμασία ήταν πάρα πολύ σημαντική για να κατανοήσει κανείς το πλήρες εύρος του, της δέσμης. Δύο χρόνια περίπου μας πήρε η προετοιμασία τις δέσμες. Μερικές φορές ξέρω ότι δείξατε σημάδια ανυπομονησίας, αλλά πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να περιμένουμε, άξιζε το, άξιζε τον κόπο όλες αυτές οι συνεδριάσεις, ε, οι ε, ατέργαστήρια, ε, οι συναντήσεις με τους εμπλεκομένους, έτσι ώστε η δέσμη να είναι σωστή. Είμαι δε απολύτως πεπισμένη ότι στο τέλος προτείναμε κάτι εξαιρετικά ισορροπημένο. Ε, μία πρόταση η οποία πιστεύουμε ε, ή μάλλον είμαστε απολύτω πεπισμένοι ότι μπορεί να υλοποιηθεί και ε, που μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο ε, βήμα έτσι ώστε να επιτύχουμε τους πολιτικούς μας ε, στόχους που είχαμε θέσει από την αρχή. Επιτρέψτε μου τώρα να ασχοληθώ με τα ε, κύρια θέματα, τις επιμέρους παραγράφους και να αναφέρω κάποια σημεία από τον οποίο ξέρω ότι θα έχετε παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Πρώτον, κινητικότητα ανταγωνιστική και δίκαιη. Το λέω ότι η κατάσταση των πραγμάτων ε, δεν είναι, ε, το status quo δεν είναι εναλλακτική ε, αποδεκτή. Υπάρχει έλλειψη κανόνων, έλλειψη υλοποίηση και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, υπάρχει ασάφεια και υψηλότερο κόστος για την βιομηχανία και βεβαίως προκύπτουν και πολλά κοινωνικά ζητήματα τα οποία συνδέονται με το στρες των ε, οδηγών και των εργαζομένων γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε να απαντήσουμε με, ε, στα όλα αυτά τα προβλήματα με πραγματικά ευρωπαϊκή απάντηση και ελπίζω ότι θα ε, αναγνωρίσετε ότι έπρεπε να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση και επομένως ε, δεν μπορούσαμε να βρούμε μία λύση η οποία να ισχύει μόνο για ορισμένα κράτη-μέλη. Βεβαίως, βεβαίως ε, ε, ανέφερα προηγουμένως ε, τις εταιρείες letterbox, ε, τις εταιρείες οι οποίες έχουν μονάχα ταχυδρομική θηρίδα, τις ψεύτικες πλασματικές εταιρείες. Έπρεπε οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και βεβαίως και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να καταπολεμήσουν την απάτη και να σταματήσουν αυτές τις παράνομες πρακτικές. Αυτό λοιπόν που μας ε, ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζονται αυτά που σας προανέφερα. Ένα άλλο θέμα που αφορά στην ανταγωνιστικότητα και τη δικαιοσύνη έχει άμεση σχέση με το καμποτάζ. Αυτή τη στιγμή οι κανονισμοί είναι πολύ περίπλοκοι, το ακούμε αυτό από πολλά κράτη, από τον Βορρά, τον Νότο, από την Ανατολή, από τη Δύση. Όλοι λένε ότι το καμποτάζ όσο έχει σήμερα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και είναι πολύ δύσκολο και να ελέγχει κανείς την εφαρμογή του καμποτάζ. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απλουστεύσει αυτού του κανόνες. Υπάρχει ένα νέο όριο των πέντε ημερών που προτείνουμε και απεριόριστο αριθμό δράσεων μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο. Αυτό όμως ε, δεν θα προσφέρει ούτε το άνοιγμα ούτε το κλείσιμο της αγοράς και εμείς αυτό επιθυμούσαμε. Σας καλώ λοιπόν να μην κρίνετε την πρωτοβουλία κάτω από αυτό το πρίσμα αλλά κάτω από το πρίσμα της απλούστευσης και της εφαρμογής των κανόνων. Αυτό ήταν το κίνητρό μας ε, και ελπίζω η πρότασή μας να είναι αρκετά ισορροπημένη για να μπορεί και να γίνει αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, ο έλεγχος των εθνικών αρχών θα είναι πλέον πολύ πιο εύκολος και Λόγω αυτού θα περιοριστεί και το παράνομο καμποτάζ, παράνομες δράσεις καμποτάζ. Όσον αφορά τώρα την ε, εφαρμογή της οδηγίας περί απόσπασης εργαζομένων στον τομέα των ε, οδικών μεταφορών, εμείς πάντα λέγαμε ότι θα πρέπει να ισχύει αυτή η οδηγία στον τομέα των μεταφορών. Το γεγονός ε, ότι οι εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα κινητικοί θα δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξερούνται από τα ωφέλη της ενωσιακής νομοθεσίας. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και πάλι να εξευρεθούν ευρωπαϊκοί κανόνες για αυτό το θέμα. Προτείνουμε το εξή να μειωθεί το ε, διοικητικό φορτίο, το διοικητικό βάρος ε, για οδηγούς ε, φορτηγών διότι μερικοί ισχυρίζονται ότι εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Δεύτερον, να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν πιο αποτελεσματικά μέτρα σε αυτόν τον τομέα. Παραδείγματο χάρη ψηφιακή ταχογράφη, ηλεκτρονικά σημειώματα παράδοση, Αυτά στο μέλλον μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες. Και όπως θα σας δείξω και αργότερα, θα πλουστευτούν οι διαδικασίε. Τρίτον, να υπάρχει ένα κατόφλι για την εφαρμογή του ελάχιστου κατώτατου μισθού. Σήμερα η οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων δεν διευκρινίζει πώς να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας. Η δική μας πρόταση είναι οι αγώνες για την ε, αποζημίωση των εργαζομένων θα ισχύουν στους οδηγούς μετά από τρεις μέρες κάθε μήνα που έχουν εσωρευτεί σε ένα κράτος μέλος. Να σας πω με απόλυτη σαφήνεια ότι σήμερα μιλάμε για το απόλυτο μηδέν. Άρα δηλαδή μετακινούμε από το 0 στο 3 στις 3 ημέρες και εξηγούμε γιατί αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης να αντιμετωπιστούν απαράδεκτες κοινωνικές ε, πρακτικές όπως οι αποκαλούμενοι νομάδες οδηγοί. Θέλουμε να δίνουμε δυνατότητα στους οδηγούς να επιστρέφουν στα σπίτια τους σε τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον κάθε τρεις εβδομάδες. Επίσης οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν κατάλληλο κατάλημα μέσα στην, στο φορτηγό όταν λείπουν από το σπίτι τους και εκτός από αυτό επίσης Εξάλλου, οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν εκπεριτροπής ρυθμίσεις. Επ' αυτού του σημείου θέλω για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, να μην προτείνουμε συγκεκριμένα ωράρια και χρόνους ανάπευσης. Ε, έτσι και αλλιώ θα υπάρξει βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων, όχι όμως με αυτές τις προτάσεις. Φτάνω λοιπόν σε αυτό τώρα το δεύτερο σημείο. Φτάνω στην ε, κινητικότητα, καθαρή και βιώσιμη κινητικότητα. Όπως σας είπα ήδη στην αρχή, δυστυχώς υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συμφόρηση. Και νομίζω ότι πρέπει να σας αναφέρω ότι εμείς μιλάμε για περίπου ένα δισεκατομμύριο την ημέρα για να αντιμετωπίσετε η συμφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και λόγω του θορύβου έχουμε υπολογίσει ότι πάνω από 100 δις ευρώ δαπανώνει το χρόνο για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Πολύ σοβαρό το πρόβλημα και προβλέπεται μάλιστα και ότι θα επιταθεί περαιτέρω κυρίως στις οδικές μεταφορές. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Με την αναθεώρηση της οδηγίας για την Ευρωβινιέτα, εμείς προτείνουμε να είναι σαφής η τιμολόγηση έτσι ώστε να χρησιμοποιείται η υποδομή πιο αποτελεσματικά. Επίσης, να επιβραβεύεται η χρήση καθαρών οχημάτων. Οι κανόνες τιμολόγησης δεν θα πρέπει να ισχύουν μόνο στα αυτοκίνητα αλλά και τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τα λεωφορεία θα πρέπει και αυτά να καλύπτονται από την οδηγία γιατί και αυτά συμβάλλουν στην εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Άρα δηλαδή αντιμετωπίζουμε στη ρίζα και στην πηγή όλες, ε, όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Βεβαίως τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν μόνα τους κατά πόσον η πρόσβαση στην υποδομή θα χρεώνεται ή όχι. Εάν όμως εισαχθούν ε, τέλη για τη χρήση των οδών, δεν θα πρέπει να βασίζονται στο χρόνο όπως αναφέρθηκε στο, αναφέρθηκε στο τελευταίο ψήφισμα που εγκρίθηκε και από το Κοινοβούλιο. Και αυτό θα πρέπει να έχει σχέση και με την αποτελεσματικότητα και με την δικαιοσύνη, γιατί η απόσταση είναι ένα καθαρό, ένα ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη προϋπόθεση και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα. Ε, το λέω αυτό ε, διότι υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία ε, έχουν προβινιέτες που τις χρησιμοποιούν και για την κοστολόγηση χρησιμοποιείται το παλιό σύστημα. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι ε, ε, οι υπηρεσίες που προσφέρονται με ΦΠΑ, με ΦΠΑ αυτές ε, οι υπηρεσίες προβλέπουν την ελάχιστη τιμολόγηση κυρίως όταν η αυτόνομη οδήγηση επικρατεί όλο και πιο πολύ το εξωτερικό κόστος και η εξωτερική τιμολόγηση είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να επιβραβεύσουμε καλύτερα τα καθαρά οχήματα. Προτείνουμε να το κάνουμε αυτό με την τροποποίηση του κανονισμού περί του του άνθρακα, γιατί το 75% ισχύει για όλα τα οχήματα που εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα και όπως σας είπα και προηγουμένως αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις κοινωνικο-οικονομικές που αντιμετωπίζουμε. Φτάνω λοιπόν στο τρίτο σημείο, στην, ε, στη συνδυασμένη κινητικότητα. Ε, νομίζω ότι η ψηφιοποίηση είναι καθοριστική σημασία για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Δεν μπορούν να είναι εμβαλωματικές οι ρυθμίσεις, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, εφόσον υπάρχουν διασυνοριακές μεταφορές. Η Κομισιόν προτείνει νέους κανόνες που θα ε, προβλέπουν ε, μία μονάδα, ένα συμβόλαιο, ένα τιμολόγιο. Αυτό θα διευκολύνει τις μεταφορικές εταιρείε και τους μεμονωμένους χρήστες των οδικών μεταφορών. Βλέπουμε εδώ να υπάρχουν και ομοιότητε με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ένας άλλος βασικός τομέας όπου προτείνουμε περαιτέρω την ψηφιοποίηση είναι την ε, χρησιμοποίηση των, αγών, των κανόν της αγοράς. Ε, αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη δεν έχουμε πολλές δυνατότητε να επιβάλλουμε αυτούς τους κανόνες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχουν σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία έτσι ώστε η έλεγχη να είναι πιο αποτελεσματική και πιο στοχευμένη. Εμείς προτείνουμε τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα την ηλεκτρονικά σημειώματα παράδοσης που αναγκάζουν ε, τις εθνικές αρχές ε, να τα αναγνωρίζουν. Θέλουμε επίσης ε, να επεκταθούν περαιτέρω οι ψηφιακοί ταχογράφοι, λιγότερη έλεγχοι σε εκείνους τους παρόχους που προσπαθούν προσπαθούν να εφαρμόσουν, να εισάγουν τέτοιου ταχογράφου Και προτείνουμε και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη από, ανάμεσα στις ε, τράπεζες δεδομένων, όπως είναι η ERRU, άρα δηλαδή ε, με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να προσφέρονται ακόμα περισσότερα δεδομένα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα μέτρα θα προτείνουν την γραφειοκρατία σε ένα τομέα που αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να υπάρχουν απλουστευμένοι έλεγχοι. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι έχουμε επιτάπητος ένα πολύ σημαντικό πακέτο, μια δέσμη μέτρων που θα έχει επιπτώσεις. Ξέρω ότι σας απασχολούν όλα αυτά, γι' αυτό και εγώ ελπίζω ότι ότι έγκαιρα θα μπορούμε να εξετάσουμε τη δέσμη μέτρων και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής μας θητείας. Είμαστε εδώ, θα κάνουμε ό,τι θέλετε να κάνουμε έτσι ώστε και εμείς ε, ε, να μπορούμε να αποκτήσουμε τις ε, απαραίτητες πληροφορίες για να προχωρήσουμε όσο πιο εύκολα γίνεται. Ναι. ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Είναι βέβαια πάντα περιορισμένος ο χρόνος. Αρχίστε εσείς, κύριε Βιμ Βάντε Κάμπ. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε. Έχω ορισμένε συγκεκριμένες ερωτήσεις που ελπίζω θα μπορέσει να απαντήσει η κυρία Επίτροπος. Σύντομα. Εμεί η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, θα, θα εξετάσουμε προσεκτικά τι προτάσει σα. Διότι υπάρχουν αρκετά καυτά θέματα μεταξύ αυτών. Και πρώτο, ο σχεδιασμός. Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω, έχουμε την πρόθεση να έχουμε ολοκληρώσει την εξέτασή τη μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Αλλά τι γίνεται με το Συμβούλιο. Αυτό ήταν το πινκ τώρα περιμένω το δικό σας pong. Όπως είπα πριν, άρχισε αμέσως το Συμβούλιο. Έχουν προβλέψει 24 συναντήσεις φέτος και πρόκειται να υποβάλουν την πρώτη ας πούμε, πρόταση φέτος τον Νοέμβρη στο Συμβούλιο. Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Βαντεκάμπ. Το σημειώνω ε, επίσης, η ερώτηση τώρα για το καμποτάζ. Περνάτε πλέον από τα λόγια στα έργα. Τρεις δράσεις σε επτά ημέρες. Και τώρα προχωρείτε σε πέντε ημέρες απεριόριστο καμποτάζ. Ναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα του καμποτάζ μέχρι σήμερα ήταν ότι αυτές, αυτές οι τρεις δάσεις σε 7 ημέρες ήταν αδύνατο να πετύχουν. Και αυτές είναι οι προφορίες που λαμβάνουμε από τον ίδιο το χώρο. Οι προφορίες που μας δίνουν τα διάφορα Υπουργεία άμεσα σε μένα και εγώ στο Συμβούλιο. Αναζητούμε δύση λοιπόν που ούτε θα ανοίξει ούτε θα κλείσει την αγορά αλλά που ταυτόχρονα θα επιτρέψει την εφαρμογή δηλαδή το χρονικό πλαίσιο που να είναι ευκολότερο να ελεγχθεί, διότι αυτές οι δράσεις ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν. Γι' αυτό προτείνουμε τώρα τις πέντε ημέρες, που είναι και ουδέτερες, δηλαδή ούτε ανοίγουν ούτε κλείνουν την αγορά. Ο κύριος Βαντικάμπ, αντιλαμβάνεστε ότι εάν είναι πέντε ημέρες σε μια χώρα, μπορεί να είναι μια μεγάλη αλυσίδα επιχειρήσεων, ε, δηλαδή δράσεων καμποτάζ. Πώς θα αντιμετωπίσετε την υπόθεση αυτή του ελάχιστου μισθού από την πρώτη μέρα και ποια είναι η εγγύηση ότι θα πετύχει αυτό. Απάντηση. Πρώτα πρώτα, από το πρώτο λεπτό της δράσης καμποτάζ ισχύει η οδηγία απόσπαση εργαζομένων. Posting. Αρχίζει αμέσως να λειτουργεί, να ισχύει η οδηγία. Καλώς συνεχίζει με τις ερωτήσεις ο κ. Βαντεκάμπ. Γιατί χρειάστηκε τόσο πολύ για τη χρήση των εφιών ταχυγράφων. Απάντηση, εγώ κληρονόμησα τον φάκελο αυτό και ανεζήτησα άλλη λύση. Γι' αυτό προτείνω κίνητρα εγώ θεωρώ ότι όλα τα εμπορικά οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν το νέο ψηφιακό ταχυγράφο ή ταχογράφο. Αλλά επίσης αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι που λέει, η νομοθεσία που λέει ότι όλα τα νέα φορτηγά θα πρέπει να έχουν τον νέο ψηφιακό ταχογράφο από το 2019. Και τα κίνητρα που έχουμε περιλάβει στο πακέτο ε, θα σας επιτρέπουν να έχετε λιγότερους συνοριακούς ελέγχους και επομένω όλο και περισσότερες υπηρεσίες και επομένω όλο και περισσότερε εταιρείε θα θέλουν να βάλουν το νέο ταχογράφο και σε παλαιότερα φορτηγά αυτοκίνητα. Μάλιστα. Θα τα περιλάβουμε αυτά σε τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάντε Κάμπ για την ομάδα των σοσιαλιστών. Θα δώσω τον λόγο σε ποιον σε εσά κυρία μου για το πινκ με την Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπο που ήρθατε ενώπιόν μας ε, και πιστεύω ότι θα συζητούμε συχνά για τα θέματα που μας απασχολούν. Ε, συνέχιση των ερωτήσεων ε, του κύριου Βοντενκάπ για τον έλεγχο. Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα, θα αυξήσετε ε, τον αριθμό των ε, ε, σημείων του καμποτάζ χωρίς όμως να υπάρξουν αδικίες ή παρανομίες. Πώς είσαστε σίγουροι ότι δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των απατών. Well, uh, απάντηση. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι ε, αδύνατο να ελέγξει κανείς τις ίδιες τις δραστηριότητες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, αντιστρέψαμε κατά κάποιο τρόπο την λογική του ελέγχου. Ε, και ε, αποφασίσαμε να δούμε το χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή ε, στο πενθήμερο καμποτάζ δεν αναφέρει μονάχα, αναφέρεται μονάχα σε μία χώρα αλλά και σε γειτονικέ χώρες όταν μιλάμε για μικρές χώρες. Επομένως καμποτάζ και με τις γειτονικέ χώρες. Είμαι σίγουρη ότι και μέσα από την βοήθεια που θα μας δώσουν οι ψηφιακοί ταχογράφοι θα μπορέσουμε να ε, ε, βρούμε λύση. Βεβαίως ε, ενθαρρύνουμε και τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν σωστές τράπεζες δεδομένων, βάσεις δεδομένων, έτσι ώστε να γίνεται και η καλή ανταλλαγή των στοιχείων. Χρειάζεται λοιπόν ε, καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών. Ε, άλλη ερώτηση όσον αφορά τους ε, ταχυγράφους. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μια ημερομηνία πιο κοντινή από, το, αυτή που προτείνεται, πιστεύετε ότι αυτό το στοιχείο ελέγχου και προστασίας θα μπορέσετε, προστασίας των οδηγών θα το στηρίξετε απάντηση. Ε, βεβαίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα είμαστε παραπάνω από ευτυχεί αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε ε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην ε, πρόταση. Το κόστος ε, του ταχογράφου λαμβάνεται υπόψη. Εάν διευρύνουμε τον αριθμό των χρηστών, σίγουρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά θα έχουμε τις θεσμικέ πληροφορίε έτσι ώστε να μπορέσουμε να, με μεγαλύτερη ασφάλεια να απαντήσουμε περί το τέλος του έτους. Άλλη ερώτηση. Όσον αφορά οχήματα κάτω των 3,5 τόνων, ε, δεν αναφέρονται ε, ε, τα οχήματα αυτά για τις ώρες ανάπαυσης. Γιατί ισχύει αυτό. Ε, και η Γαλλία αλλά και άλλα ε, μέρη υπάρχουν πολλές χώρες λοιπόν οι οποίες ε, όντως προβληματίζονται για τα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων χρειάζεται γενικός έλεγχος γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε να προσθέσουμε την έδρα το σημείο εγκατάστασης δηλαδή αλλά πιστεύουμε ότι δοθήσεις της καταστάσεως ε, σε αυτή τη φάση για τα μικρά ε, οχήματα ε, κάτι τέτοιο υποχρεωτικό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Ευχαριστώ πολύ ο Ζήλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. πράγματι είναι λίγο σαν δικαστήριο, ναι, όχι, ναι, όχι απαντήσεις. Τέλος πάντων, είπατε ότι λάβατε υπόψη σας ε, την επιτυχία της ενεργειακής πολιτικής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όσον αφορά το αέριο. Επίσης, ε, αναφερθήκατε στο πακέτο κινητικότητας ε, για τις οδικές μεταφορές. Εκεί αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η κύρια χώρα δραστηριοποίησης ε, μιας εταιρείας. Ε, κατ' ουσίαν τι θα κάνουμε, θα ακολουθήσουμε μια κατεύθυνση και στις αεροπορικέ μεταφορές, στις θαλάσσιες μεταφορές, γιατί έχουμε πολλά κράτη-μέλη που στις ταχυδρομικές υπηρεσίες αναπτύσσουν δραστηριότητα σε άλλο κράτος ε, μέλος. Δηλαδή αυτά που είπατε περιούνται μόνο σε οδικές μεταφορές. Κοιτάξτε, η δέσμη μέτρων αφορά εγώ αναφέρομαι όχι στην δέσμη μέτρων, αναφέρομαι στην φιλοσοφία, τη γενικότερη. Ε, δηλαδή θα έχει κανείς μια κύρια χώρα που αναπτύσσει δραστηριότητε, θα ισχύσει αυτό και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε την προσοχή μας στις οδικές μεταφορές, αλλά όπως ε, είδατε έχουμε καταβάλει πολλές ε, προσπάθειες για να υπάρχουν ε, ίσοι όροι ανταγωνισμού και αυτό που θα κάνουμε είναι θα εξετάσουμε καλύτερα τις κοινωνικές πτυχές της αεροπλοείας στο τέλος του έτους και θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε ποιος ε, θα πρέπει και ποιος θα είναι ο κοινό παρονομαστής για όλα τα μέσα μεταφοράς, έτσι ώστε να ισχύουν παντού τα ίδια. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε επίσης ε, ε, να μπορεί να πηγαίνει ο εργαζόμενος μετά από τρεις ε, εβδομάδες στο σπίτι του. Σπίτι του τι είναι, εκεί που ζει ή εκεί που είναι η εταιρεία του. Αν αναφέρεται στη διέσβη μεταφορών, σπίτι είναι εκεί όπου ε, έχει την έδρα της εταιρεία. Αλλά ο οδηγός και τα φορτηγά ε, μπορούν βεβαίω να κυκλοφορούν ε, χωρίς περιορισμό ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές ε, του φορτηγού. Το φορτηγό δεν πρέπει να γυρίσει πίσω. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας μπορεί να αλλάξει τον οδηγό. Άλλο ρώτησα εκεί που είναι καταγεγραμμένη η εταιρεία του είναι το σπίτι ή η ηθαγένειά του. Γιατί στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ελεύθερη μετακίνηση. Μπορεί και να ζει σε άλλη χώρα μόνιμα από αυτήν στην οποία εργάζεται. Ε, λυπάμαι εδώ, δεν μπορώ να απαντήσω. Ε, μάλλον έπρεπε να ρωτήσω και μου είπαν εκεί που είναι επίσημα καταγεγραμμένος ο οδηγός, όχι δηλαδή η εταιρεία του. Όσον αφορά τώρα τα κοινωνικά θέματα, ε, κατανοώ ότι είναι δύσκολο να υπάρχει συμβιβασμό. Ο Ρουμάνος αισθάνεται καλύτερα να ε, κοιμάται στο φορτηγό του ε, και να μην κινδυνεύει το φορτίο του γιατί μπορεί κάτι να συμβεί και μετά να χάσει ε, τη δουλειά του στη Ρουμανία. Ε, πού ε, είναι πιο ασφαλής, το να κοιμάται μέσα στο φαρτηγό ή το να είναι άνεργο στη Ρουμανία. Είμαι σίγουρο ότι αυτό θα συζητηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Κοιτάξτε, αν δείτε λιγάκι ε, αν δει κανεί το συμβιβασμό που πετύχατε, ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ερωτώ ε, σε γενικές γραμμές πόσο είσαστε ικανοποιημένοι σχετικά με αυτή τη δέσμη μέτρων. Κυρίως ε, έχοντας κατά νου την κοινή αγορά, είσαστε ικανοποιημένοι κατά 60, 70, 80%. Κοιτάξτε, δεν είναι δικό μου, δεν είναι δική μου αυτή η δέσμη μέτρων. Είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους. Εγώ πιστεύω ότι καταθέσαμε μια πολύ ισορροπημένη πρόταση και βέβαια σε ορισμένα θέματα έχουμε διαφορετική άποψη διαφορετικές ομάδες άμεσα ενδιαφερομένων, αλλά είμαι πεπισμένη ότι τελικά ε, θα πλησιάσουμε. Ε, θα είναι καλή η πρόταση Κομισιόν, γιατί είναι ισορροπημένη. Και λάβαμε υπόψη μας πρώτα απ' όλα τον, την Ευρωπαϊκή Συνθήκη που λέει ότι το άνοιγμα της αγοράς θα πρέπει να γίνεται σταδιακά, να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες στα κράτη-μέλη και δεύτερον, ο στόχος αυτής της δέσμης μέτρων δεν αφορά τόσο το άνοιγμα ή το κλείσιμο της αγοράς, αλλά αφορά στην διευκρίνηση κανόνων που έχουν σχέση και με τη νέα τεχνολογία, άρα δηλαδή ε, να υπάρχει διαφάνεια. Ε, τώρα ε, στους, στις οδικές μεταφορές επικρατεί χάος και πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για να υπάρξουν καλές συζητήσεις στο μέλλον. Άρα δηλαδή η διευκρίνηση ενός πράγματος που θα είναι διαφανές και βέβαια μετά ανάλογα με τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη, θα ακολουθήσουν και άλλες συζητήσεις. Υπενθυμίζω λέει η Πρόεδρος ότι προφανώς δεν πρόκειται για δικαστήριο δεν έχουμε ε, ακρόαση, επακροατήριο εδώ πέρα. Δεν ε, κάνουμε συζητήσεις. Την επόμενη φορά, ε, για να είμαστε όλοι χαλαροί και ωραίοι, θα φέρω και λίγο κρασάκι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση, γιατί το θέμα μας είναι να συζητήσουμε, να προωθήσουμε το θέμα επί της ουσίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι θέλουμε όχι απλά αποσαφηνήσει. Ε, ε, εγώ προσδοκώ να ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ελεύθερη αγορά, την εσωτερική αγορά να την ολοκληρώσουμε, να την εμβαθύνουμε και όχι απλά να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτό το ξεκαθαρίζω εξ αρχής. Μιλήσατε για την ε, ενιαία αγορά, μετά μιλήσατε για κάτι το οποίο υφίσταται σήμερα στην αγορά, ε, ε, που είναι ο προστατευτισμός και που δεν είναι παράτυπη ή αθέμητη πρακτική. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι αν υπάρχει ισορροπία. Ίσως στο τέλος να έχουμε ισορροπία, αλλά οι δύο ανασχετικές μειοψηφίες στο Συμβούλιο έχουν στη μέση τους κάποιες ε, χώρες οι οποίες ε, ε, μετακινήθηκαν νομίζω κάποια στιγμή προς την ανασχετική μειοψηφία. Τι γίνεται όσον αφορά την εσωτερική αγορά, ποια είναι τα μέτρα κύριε Επίτροπε. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία πιστεύετε ότι θα οικοδομήσουν, θα σφυρατήσουν καλύτερα την εσωτερική αγορά. Κοιτάξτε, η διευκρίνηση αφορά όχι ολόκληρη την δέσμη, αλλά το καμποτάζ. Ε, αυτό που θέλησαμε να κάνουμε στο καμποτάζ είναι να διευκρινίσουμε τους κανόνες. Ένα άλλο, ε, ε, μεγάλο, μια μεγάλη μεγάλη βελτίωση που είναι σίγουρα βελτίωση κατά 100% αφορά την ψηφιοποίηση. Όλα τα, έχουμε τέσσερα μέτρα που αφορούν την ψηφιοποίηση και που θα μειώσουν το ε, άχθος, το διοικητικό και, την, και επομένως θα βελτιώσουν πολύ την κατάσταση. Να σας πω κάτι που με σοκάρισε. Είναι γεγονός ότι με 28 χώρες μέλη, 27 25 ε, χώρες μέλη δεν χρησιμοποιούν σωστά το ε, κεκτημένο ε, και είναι και πολλές αυτές οι οποίες το εφαρμόζουν μεν αλλά όχι με τον ανάλογο τρόπο. Επομένως με την πρόταση αυτή έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ε, μιλάμε λοιπόν για ψηφιοποίηση, μιλάμε για την μείωση του, των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος. Ε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει και ο χρήστης πληρώνει. Ξεκαθαρίστηκαν κάποια πράγματα γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε η Κομισιόν να τα κάνει γιατί δεν είχε στη διάθεσή της ε, ψηφιακά εργαλεία. Ε, στην ουσία δηλαδή η Κομισιόν κάνει αυτά που τη ζητούσε ο τομέας εδώ και πάρα πολύ ε, καιρό, ότι ο Ριπένον πληρώνει. Είμαι πεπισμένη ότι με πολλαπλούς τρόπους αποτελεί βήμα προς, προς τα εμπρός αυτό, αυτή η δέσμη. Ε, τώρα το άνοιγμα της αγοράς δεν ήταν στόχος ε, του πακέτου. Ε, ε, η δέσμη αυτή έχει σαν στόχο να θέσει σαφείς κανόνες και βεβαίως όπως είπα και από την αρχή πολύ περισσότερη δουλειά θα γίνει στο μέλλον. Εγώ αναφερόμουν στην ε, καλύτερη λειτουργία της ε, ε, αγοράς. Δεν αναφερόμουν μόνο στην ψηφιοποίηση κτλ. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι ψεύτικες, είναι letterbox μόνο. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες για αυτές, να ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες για το καμποτάζ, ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες για την οδηγία ε, των ε, αποσπασμένων εργαζόμενων και αναφερόμαστε σε τρεις μέρες για τους οδηγούς διεθνών μεταφορών. Γιατί αυτό είναι λογικό. Από τη στιγμή που απλώς παραλαμβάνει, συγγνώμη, δίνεις εμπορεύματα, σε εμπορεύματα δεν εμπίπτει ε, στους ε, ε, αποσπασμένους εργαζόμενους από τη στιγμή που ξαναφορτώνεις τότε υπόκειζε στην νομοθεσία αυτή. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και οπωσδήποτε στο μέλλον θα το κάνουμε. Ίσως έθεσα λάθος ερώτηση. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο εστιασμένος σε συγκεκριμένα θέματα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενίσκα. Η κυρία Κέλλενεν για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που ήρθατε καταρχήν στην Επιτροπή μας και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο και δύο ερωτήσεις. Έχουμε πάρα πολλούς ε, κανισμούς. Ε, ε, υπάρχουν κανισμοί που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη και δεν υπάρχει έλεγχος, ούτε επιβάλλονται και κυρώσεις. Αυτό λοιπόν το γεγονός στρεβλώνει την αγορά της, των μεταφορών στην Ευρώπη. Και ερωτώ, πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να αποφύγουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στο Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση ακριβώς σε αυτό το θέμα. Και ποια είναι η άποψή σας, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το πολυτροπικό σύστημα μεταφορών, να βελτιώσουμε το, τις υποδομές, ε, τα λιμάνια, τους σιδηροδρόμους. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση σχετικά με την ε, συνεργασία και την ε, εφαρμογή των κανόνων, αυτό μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη διαφάνεια και με το να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες στην Εθνική Τράπεζα Δεδομένων, όπως την ERRU, στο Ευρωπαϊκό Μητρό Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών. Εκεί μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία των κρατών μελών ε, και μπορούμε και να επιβάλλουμε την εφαρμογή αν δεν το πράττουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, σε τελική ανάλυση, η μη συνεργασία μπορεί και να στοιχήσει και την άδεια σε μια εταιρεία, αν δηλαδή η εταιρεία δεν σέβεται το κοινοτικό κεκτημένο. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά τώρα την πολυτροπικότητα, ε, εμείς ε, εφαρμόζουμε και αυτά που προτείνει το Κοινοβούλιο, δηλαδή σωστή τιμολόγηση, στην τιμολόγηση να λαμβάνουν υπόψη και εξωτερικοί παράγοντες. Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Δηλαδή έχουμε εισαγάγει την αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει και ο χρήστης πληρώνει και όχι μόνο αυτό, αλλά η νέα μέθοδος τιμολόγησης δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να επιβάλλουν τέλη συμφόρησης, ε, τέλη δηλαδή αν υπάρχει ένας τομέας που είναι ιδιαίτερα, που υποφέρει από τη ρήπανση, εκεί μπορούν να επιβληθούν ειδικά τέλη για να μειωθεί η ρήπανση αυτή τη συγκεκριμένη περιοχής. Και το και για τη συμφόρηση. Αν έχουμε μια περιοχή με μόνιμη συμφόρηση, ε, υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες, τρόποι για να περιορίσει κανείς τη συμφόρηση. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι ε, δυνατότητες και νομίζω ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά να ε, φτάσουμε στο να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα στη χρήση των ε, διαφόρων μέσων μεταφοράς. Εγώ ρώτησα πώς θα αποφύγουμε τη σύγκρουση Βορρά, Νότου, Ανατολής και Δύσης. Ε, επ' αυτού του θέματος. Και εγώ να ρωτήσω πόσο χρόνο έχω για να απαντήσω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Ένα πράγμα είναι απόλυτα σαφές. Τα θέματα που έχουν τεθεί επιτάπητο, κατά την άποψή μου δεν αφορούν τη σύγκρουση βορρά-νότου-ανατολή Δύσης. δυση ειναι θέματα μεταφορών. Αφορούν το, τις μεταφορές ε, του μέλλοντος. Ενιαίος χώρος μεταφορών, ενιαία αγορά. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Και εγώ ε, τα έχω μόνιμα κατά νου για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το ε, πώς ε, η νομοθεσία μας, η δουλειά μας επηρεάζει το κόστος ε, της λειτουργίας και επηρεάζει και την κινητικότητα των ανθρώπων. Έτσι μόνο κατανοεί κανεί τη σημασία της νομοθεσίας. Δεν πρόκειται για τη σύγκρουση βορρά-νότου, ανατολής-δύσης. Το θέμα είναι να παραμείνει ανταγωνιστική αγορά, να υπάρξει σταδιακά η, η επίτευξη η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς. Άρα δηλαδή ε, πρέπει να κάνουμε τα βήματα σιγά σιγά, αυτή είναι η μόνη λύση. Τα μικρά σταθερά βήματα οδηγούν σε μεγάλες αλλαγές. Αυτά όμως ε, πρέπει να γίνονται και με ένα συνετό τρόπο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί ξέρετε το όλο θέμα έχει και καθαρά πολιτική χρειά. Ε, πρέπει να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας, να κατανοήσουμε ότι για να συμμετάσχει κανείς πλήρως σε ένα τομέα πρέπει να ανοίξει ο τομέας αυτός, αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι ιδιαίτερα αναπτυγμένοι τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, όταν ανοίγει κανείς τους οριζοντές του, τα μικρά βήματα την χάνουν αναγνώρισης και μπορεί να συνεχίσει κανείς σε μια κατεύθυνση που τελικά όλοι τη θέλουν να εφαρμόζεται πλήρως η ενιαία αγορά. Αλλά σας είπα, τα μικρά βήματα θα μας οδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Κράμερ, ο ταχογράφος είναι η λύση στην ψηφιακή εποχή, διότι και εξοικονομείται χρήματα και οι έλεγχοι είναι ε, σκόπιμοι, γιατί να περιμένουμε να εισαχθούν οι νέοι ταχογράφοι του 2019. Αυτό βέβαια το κατανοώ, αλλά γιατί δεν μπορεί να γίνει σε δύο-τρία χρόνια ο εξοπλισμό και των παλαιών οχημάτων με, ηλεκτρονικούς, με ψηφιακού ταχογράφου για να αποφευθεί και όλη αυτή, η όλη αυτή η υπόθεση με το καμποτάζ. Γιατί δεν το κάνετε. Απάντηση της Επιτρόπου κυρίας Μπούλκ. Να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, αλλά ξεκίνησε αυτό το Μάρτιο 2016 και πρόκειται να γίνει το 2019. Ε, πρόκειται για, την για τον εκ εξοπλισμό. Ναι, αλλά γι' αυτό προτείναμε κίνητρα. Πολύ ευχαρίστω να σα υποστηρίξω, συνεχίζει η Επίτροπο Συμπολούκου, για την αλλαγή του τμήματο αυτού τη προτάσεω. Σα ευχαριστώ για την απάντησή σα, λέει ο κ. Κράμερ. Δεύτερο, αθέμητο ανταγωνισμό. Γνωρίζετε τη θέση μου. 100% του σιδηροδρόμου πλέον ιδιώδια, 1% των ε, ε, δρόμων. Και τώρα λέτε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουν μειώσει 25% για τα διόδια. Θα κάνετε τα ίδια και, και για είδη ε, τρένων τα οποία πληρώνουν χρησιμοποιούν άλλα είδη ενέργειας. Κοιτάξτε, ναι, οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο μέρος των, των στην Ευρώπη είναι ήδη ηλεκτροδοτημένοι γινόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση των δυνατών συντόματων, αλλά πολύ συχνά λέμε σιδηρόδρομος και οδικές μεταφορές είναι υπορισμένες συνθήκες τα ίδια. Όχι, πρέπει να μιλούμε για σιδηροδρόμους, αλλά ο σιδηρόδρομος έχει περιορισμένη ακτίνα δράσος. Ο δρόμος πηγαίνει πολύ μακρύτερα και έχουμε και όλα τα ενδεχόμενα ε, επίπεδα απατών και ταυτόχρονα υπάρχει και ανταγωνισμός για τον σιδηρόδρομο. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτή την έλλειψη ισορροπίας στην προσέγγιση όπου και αν εντοπίζεται αυτή. Και θα είδατε κι εσείς, Μικαέλ, και με όλη τη δουλειά που έχετε κάνει, ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό τώρα με τρόπο συστηματικό. Και μπορώ να σας πω επίσης ότι σχεδιάζουμε να κάνουμε και άλλα, να λάβουμε και άλλα μέτρα για την sharing economy και τις μεταφορές με το σιδηρόδρομο συνεργαζόμενοι ταυτόχρονα και με άλλους ε, επιτρόπους για να κλείσουμε τον κύκλο, διότι δεν είναι μονάχα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι και η καθαρή ενέργεια και η ενέργεια που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα. Πρόκειται για συνεργασία, δηλαδή μπορούμε να πάμε και γρηγορότερα, μάλλον μπορούμε. Αλλά ας αναζητήσουμε τον καλύτερο τρόπο πώς να το κάνουμε χωρίς να προκαλέσουμε καταστροφές. Να συνεχίσουμε δηλαδή την εξέλιξη. 100% ηλεκτροδοτημένοι ε, σιδηρόδρομοι είναι μόνο στην Ελβετία. Αυτό είχε ήδη εγκριθεί στη Γερμανία προ 110 ετών και ακόμα βρίσκεται στο 70%. Τώρα, το, το καταποκοπήν ποσό λέει η Εφατσέτ ότι το έχει δεχθεί ο Ντομπριντ. Λέει όμως τώρα ότι δεν δέχτηκε τίποτα. Ποιος λέει ψέματα εσείς ή ο Ντόμπριντ σχετικά με τα διόδια των φορτηγών στους αυτοκινητοδρόμους. δεν ξέρω πώς χώθηκε και ο Αλεξάνδρ Ντόμπριντ εδώ, ο Γερμανός υπουργό. Αυτό προτείναμε εμείς είναι σαφές. Δηλαδή οι τέλη πληρώνονται στη βάση της απόσταση διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποκλείσουμε τα εξωτερικά στοιχεία. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει καμία ξεκάθαρη θέση. Έχουμε κάποιες διασφαλίσεις από χώρε που έχουν ήδη την Ευρωβινιέτα, δηλαδή ε, ε, ε, ποινιέτες που πληρώνονται ανά έτος, έχουμε επιχειρήματα που λένε ότι αυτό απλώς σημαίνει μια μεταβατική περίοδο. Και το distance-based charging θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε αν είχαμε τη σχετική τεχνολογία. Δεν την έχουμε. Τώρα που προχωρεί τόσο ταχύτατα η ε, ψηφιοποίηση, μπορούμε να το κάνουμε ως επόμενο βήμα. Λούντγκριν, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα έχω να τονίσω κάποια πράγματα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η φυστάμενη νομοθεσία. Όχι. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ε, για επτά ε, ημέρες τρεις δράσεις. Και εκεί ήταν ακριβώς το παραθυράκι. Αν υπήρχε μία φράση που να έλεγε ότι μετά από την χρήση μιας περίοδου καμποτάζ μέσα στην χώρα προορισμού το φορτηγό θα πρέπει να επανέλθει στη χώρα προέλευσης, τότε θα είχατε λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα πλέον. Αυτό όμως που κάνατε τώρα με τη νέα πρόταση, εγώ ήλπιζα να διορθώσετε το πρόβλημα, όχι να προκαλέσετε νέα προβλήματα. Αυτό που κάνατε τώρα είναι ότι μετακινήσατε το πρόβλημα για, από εκεί που ήταν για τις μακρές διαδρομές, εκεί βρίσκουμε εμείς το πρόβλημα σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη, Σουηδία, Δανία, τους επιτρέπεται τώρα να εισέρχονται στην χώρα τη Δευτέρα το πρωί, να παραμένουν, να κάνουν απεριόριστο αριθμό μεταφορών για τη διάρκεια πέντε ημερών. Αλλάζεται, μετακινείται τον ανταγωνισμό και τον βάζετε στην τοπική διανομή. Άρα δεν είναι πλέον το πρόβλημα της αγοράς long haulage. Τώρα μπορούν να ε, δουλεύουν στην τοπική διανομή. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει κάτι τέτοιο διότι να με πιστέψετε και στη δική σας χώρα, τη Σλοβενία, θα έχετε την ίδια εμπειρία. Θα πλημμυρίσουν φορτηγά αυτοκίνητα την χώρα σας που θα δουλεύουν για τα μισά λεφτά και θα σκοτώσουν την τοπική σας αγορά, όλες τις τοπικές σας επιχειρήσεις. Και μετά θα κάτσετε να μου πείτε ότι πρέπει να σκεφτούμε ενιαία αγορά, ανοιχτή αγορά. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει σε άλλε χώρε μέλη να έρθουν να σκοτώσουν την οικονομία άλλων χωρών που προσπαθούν τέλο πάντων να ζήσουν να αξιοπρεπώς. Είναι απολύτως απίστευτο ότι σκέπτεστε να τους επιτρέψετε πέντε ημέρες απεριόριστο αριθμό δράσεων. Στην ουσία πάτε από το κακό στο χειρότερο. Δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. πρόβλημα ε, δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, προκαλείται νέα. Ε, η ερώτηση. Δεν ακούσαμε την ε, απάντηση του Ευρωβουλευτού. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα διαφωνώ μαζί σας απολύτως ότι κάναμε χειρότερες τις συνθήκες και θα σας εξηγήσω γιατί. Και θα παρακαλέσω όλους τους αξιότιμους ευρωβουλευτές να ακούσουν τι έχω να πω, διότι γνωρίζω ότι πολλοί από εσά αμφισβητείτε τα, με, τα, ίδια επιχειρήματα. Πρώτα, αυτέ τι τρει δράσει κανένα δεν μπορούσε να τι ελέγξει. Οι φορτωτικέ που είχαν οι οδηγοί μπορούσαν να τι ε, επιδείξουν ή όχι. κανένα δεν τους πίεζε να τι επιδείξουν, μπορούσαν να τι κρύψουν κατά το τραπέζι και να μην το ξεγνωρίζει κανεί ότι υπάρχουν. Απολύτω ανέλεγκτη η κατάσταση, ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Εγώ πήγα σε ελέγχου ε, που, που έκανε η τροχέα και ήταν φοβερά τα πράγματα προσπαθήσαμε με την υπηρεσία μου να φτιάξουμε κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε να λειτουργεί μέσα στο στόχο. Δηλαδή ούτε άνοιγμα ούτε κρίσιμο τη αγορά. Τώρα βεβαίω θα είναι δυνατόν να γίνει έλεγχο. Δεύτερον, δεν πιστεύω ότι τώρα θα πλημμυρίσουν φορτηγά. Διότι το καμποτάζ από την ημέρα αριθμό 1 μπαίνει αμέσω στην οδηγία απόσπαση εργαζομένων. Άρα το κόστο θα παίζει ρόλο στο πόσε δράσει θα κάνει μια επιχείρηση ή ένα φορτηγό αυτοκίνητο και δεν θα προκαλέσει αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν έχουμε βέβαια τόσο, δεν έχουμε περιόριστο χρόνο για να συζητήσουμε, αλλά σας προσκαλώ να συζητήσετε με τη Γενική μου Διεύθυνση, με το προσωπικό μου γραφείο, να σας τα εξηγήσουμε, γιατί προβλέπουμε πολλά στοιχεία τα οποία όλα μαζί θα προσθεθούν. Βεβαίως, και θα μπορούσαμε να κάνουμε και λάθος και βεβαίως θα υπάρχει και χώρος βελτιώσεων τους επόμενους μήνες, αλλά κάναμε τα πάντα με πραγματικά καλή πρόθεση ώστε να εξισορροπήσουμε την προσέγγιση, ούτε να ανοίξουμε ούτε να κλείσουμε την αγορά. Και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι όταν οι αστυνομικοί θα κάνουν ελέγχους, να μπορούν πραγματικά να κάνουν ελέγχους και να επιβάλλουν την εφαρμογή των κανόνων. Το καμποτάζ ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και όταν παραπονούνταν οι επιχειρήσεις, αυτό που μας έλεγαν, αυτό για το οποίο παραπονούνταν και κατήγγελαν, ήταν ότι δεν εφαρμόζονται οι κανόνες. Όταν θα εφαρμοστούν τότε θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Πιστεύω όμω ότι η πρότασή μα είναι ισορροπημένη και όντω θα εξυπηρετήσει εκείνου που χρειάζονται βοήθεια για να επιβάλλουν του κανόνε. Σαφώ δεν θα συμβεί αυτό, απαντά ο Ευρωβουλευτή. Ε, κύριε Λονγκριν, δεν έχετε άλλο χρόνο. Τέσσερα λεπτά για όλου. Το ίδιο ισχύει. Θα αφήσουμε λοιπόν του άλλου Ευρωβουλευτέ, διότι αν ο καθένα αγορεύει και δεν κάνει ερωτήσει, βέβαια αυτό είναι δικό σα θέμα. Εγώ φροντίζω να γίνει η ανταλλαγή απόψεων. Δεν έχουμε όπως είπα και ατελείωτο χρόνο. Οι υπόλοιποι τώρα ευρωβουλευτέ που λαμβάνουν το λόγο θα έχουν από ένα λεπτό. Και πρώτος ο κύριο Ντελή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο σύντομες ερωτήσει και θέλω την απάντησή σας όσον αφορά το χρόνο ανάπαυσης. Ορισμένες χώρες, όπως γνωρίζετε, έχουν πάρα πολύ ε, αυστηρούς νέους κανόνες όσον αφορά την εβδομαδιαία ανάπαυση. Θα προτείνετε ενδεχομένως ε, ε, ανέρεση των διαφόρων ε, εθνικών κανόνων που έχουν σχέση με το θέμα αυτό στη δέσμη για την κινητικότητα. Δεύτερον, το, η δέσμη αυτή της κινητικότητας θα έχει οποιαδήποτε ε, οποιαδήποτε, θα έχει οποιοδήποτε αντίκτυπο όσον αφορά τη διαδικασία επιπαραβάση που έχει ξεκινήσει η Κομισιόν ε, ε, σχετικά με τις αμοιβέ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, λέει η Πρόεδρος, και επομένως θα ακούσουμε το σύνολο των ερωτήσεων και μετά θα απαντήσει η Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας πω ότι τα λεωφορεία και τα φορτηγά δεν πετάνε. Νομίζω ότι θα πρέπει να μου πείτε το εξής. Τι γίνεται με, αυστη... Ε, με... με... Ε, ε, Ασφαλής σε χώρους ε, πάρκινγκ εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, ε, θα πρέπει να το δούμε το, το ζήτημα αυτό. Τι γίνεται. Ε, γιατί τι θα γίνει, μιλάμε για ασφαλείς μεταφορές αλλά δεν έχουμε ασφαλείς θέσεις σε πάρκινγκ. Ευχαριστώ κύριος Βαντάλεν. Έχετε εγγραφή. Μην εκπλήσεστε. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, ε, για το καμποτάζ. Είναι γεγονός ότι έχουμε προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο και σε λίγο θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο η κατάσταση. Ε, είναι οι ικανότητες πάρα πολύ μεγάλες, ε, οι έλεγχοι γίνονται μονάχα ε, σε επίπεδο τοπικής διανομής γιατί αυτές οι πέντε μέρες χωρίς κανένα άλλο όριο ή περιορισμό οπωσδήποτε θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Και οι έλεγχοι που δεν θα καταφέρουμε να να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε ούτε αργότερα να τους κάνουμε. Από τη στιγμή που δεν βελτιώνονται τα πράγματα γιατί δεν σταματάτε το καμποτάζ. Όσον αφορά τώρα ασφαλείς χώρους στάθμευσης, εγώ ε, είχα συμμετάσχει σε μία συνεδρίαση και με εκπροσώπους της Κομισιόν και υπαλλήλους λοιπά Φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο ταμείο που όλοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Επόμενη ομιλήτρια. Ε, Όσον αφορά ε, τους ε, χρόνους ανάπαυσης, θέλω να πω ότι όταν δεν υπάρχει απαραίτητη υποδομή, ποιος θα ελέγχει το αν τηρούνται οι χρόνοι ανάπαυσης ή όχι και ποιος εκτείνεται όταν έχουμε ιδιαίτερα ευπαθή εμπορεύματα Ποιος αναλαμβάνει την ασφάλισή τους. Αυτά όλα είναι σημαντικά ερωτήματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μόνο λίγους οδηγούς οι επιχειρήσεις αυτές είναι αναγκασμένες ε, να μεταφράζουν τα έγγραφα σε διάφορες γλώσσες, ε, πρέπει να κατατίθενται όλα αυτά τα έγγραφα, οι ε, συμβάσεις εργασίας. Αυτά όμως δεν οδηγούν σε απλούστευση, αλλά σε διόγκωση της γραφειοκρατίας. Και τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξαφανίσει τις εικονικές εταιρείε, αυτές που είναι εταιρείε βιτρίνας. Ε, και επίσης και μια άλλη ερώτηση. Ε, τα διάφορα συστήματα αποζημίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διαφέρουν, ε, πώς μπορείτε να τα συγκρίνετε. Και όταν κάνετε όμως τη διαίρεση δια του χρόνου εργασίας, προκύπτει, θα πρέπει να προκύπτει ο ίδιος, η ίδια αποζημίωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Πώς μπορεί κανείς ε, να επιτύχει την ε, εναρμόνιση ε, με ελέγχου, αλλά πολλές φορές οι αρμόδιοι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα του οδηγού. Πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερη, Ευρωβινιέτα. μήπω ήταν καλύτερα ότι να υπάρχει ένα στάνταρ ετήσιο ποσό. Γι' αυτό θα μπορούσε να είναι κίνητρο. Γιατί υπάρχουν κάποιες ε, οδικέ αρτηρίες ε, που πάνε παράλληλα με τους αυτοκινητόδρομους και τι κάνουν οι οδηγοί επιλέγουν αυτούς για να μην πληρώσουν διόδια. Και τέλος, όσον αφορά το καμποτάζ, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μεταφορών στις, ε, ε, στις παραμεθόριες περιοχές, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Η κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα να πω τα θετικά. Ε, χαίρομαι που επιτέλους έχει κατατεθεί αυτή η δέσμη μέτρων και θέλω να περιστώ σήμερα στην οδηγία για την Ευρωβινιέτα. Η Κομισιόν πιστεύει ότι η οδηγία αυτή και η Ευρωβινιέτα θα πρέπει να ισχύει για όλους τους τύπους αυτοκινήτων ε, διότι ε, υπάρχουν επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να προλάβουμε την διακριτική μεταχείριση. Εσείς τώρα μπορείτε να μας διευκρινίσετε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός έτσι ώστε ε, όταν πάει κανείς ιδιωτικά από το Άμστερνταμ στην Ουτρέχτη να επιβάλλεται από το κράτος ε, το τι θα πρέπει να καταβάλλεται ως τέλος ή όχι. Επίσης, ε, όσον αφορά τους φόρους για τα ιδιωτικά οχήματα, αυτό δεν αναφέρεται πουθενά παρότι προσπαθείτε να επεκτείνετε την Ευρωβινιέτα και στα ιδιωτικά οχήματα. Και τρίτον, η Ευρωβινιέτα ε, υποτίθεται θα χρηματοδοτήσει και την ε, ε, ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων και γιατί η Κομισιόν εξ αρχής δεσμεύεται για το earmarking. Τέταρτον, η Κομισιόν γιατί θεωρεί ότι συχνά μετακινούμενοι που εξαρτώνται από το αυτοκίνητο γιατί δεν έχουν άλλη δυνατότητα για να πάνε στη δουλειά τους και πολλές φορές ε, αντιμετωπίζουν και τη συμφόρηση. Αυτοί εκτός ότι κάνουν, χάνουν χρόνο να πρέπει να πληρώσουν και τέλη από πάνω. Και τέταρτον, Πόσες ε, σιδηροδρομικές ε, ενώσεις συμμετείχαν στη σύγκρουση για την Ευρωβινιέτα. Όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σμίτ. Και εγώ μια πολύ σύντομη ερώτηση. Γιατί η Ευρωβινιέτα εφαρμόζεται για τα βαρέα οχήματα, για τα φορτηγά, ενώ εγώ νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι τα φορτηγά, τα μικρά φορτηγά και τα αυτοκίνητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά την φορολογία και οπωσδήποτε να μην είναι σε εθελοντική βάση, γιατί η κλιματική αλλαγή δεν περιμένει. Ε, λοιπόν, αφήσαμε ε, περιθώριο στα κράτη-μέλη ε, και νομίζω ότι πλέον πέρασε ο χρόνος. κύριε Grass Waterheads. Και εγώ έχω μια ερώτηση για την οδηγία περί κόστους οδικών μεταφορών. Θα πω κάτι άλλο πολύ πιο σύντομο, τα οχήματα. Η Κομισιόν ανέστηλε την ε, διαδικασία. Μήπως μπορείτε να μου αναφέρετε τους πολιτικούς και τα πολιτικά και νομικά αίτια. Και υπάρχει ίσως κάποια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά τώρα το θέμα της οδηγίες περί κόστους, η Κομισιόν θέλει να εξασφαλίσει ότι για τους συχνά μετακινούμενους δεν θα προκύψει ιδιαίτερο κόστος. Κι άλλο ένα ερώτημα, μακροπρόθεσμα. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό τέλος υποδομών από τα διαφορετικά τέλη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μπαχ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για όλα αυτά που μας είπατε. Θα ήθελα να δείξω δύο θέματα. Η δεύτερη μέρα ανάπαυσης. Αυτό προκαλεί μεγάλη φασαρία. Στο Λουξεμβούργο την προηγούμενη εβδομάδα τα συνδικάτα είπαν ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη τους. Και λένε τα συνδικάτα ότι ε, επιθυμούν τον κοινωνικό διάλογο. διευθυνθεί κατεμβασίτους διαβουλευτήκατε μαζί τους ή όχι. Και δεύτερον, η έλεγχη. Η έλεγχη είναι το α και το μέγα της νομοθεσίας. Τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τους ελέγχους που είχαν υποσχεθεί. Στο μέλλον λοιπόν τα κράτη-μέλη σκοπεύετε να τους επιβάλλετε να εφαρμόζουν ελέγχους ε, και να είσαστε πιο αυστηροί. Ο κύριος Νίλσεν. Ευχαριστώ πάντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, οι κανόνες. Εάν δεν υπάρχει έλεγχος ε, εφαρμογής και αν δεν τιμωρείται ο παραβαίνουν τους κανόνες, τότε γιατί στο καλό υπάρχουν οι κανόνες. Σε γενικές γραμμές λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν καλοί, σωστοί έλεγχοι. Ναι, αλλά μήπως δεν έχουν καν προσπαθήσει τα κράτη-μέλη. Τώρα πλέον υπάρχει το κείμενο ε, και το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί σωστά και πλήρως από τα κράτη-μέλη. Ε, ε, τώρα, τι, τι θα κάνετε, κυρία Επίτροπε, έτσι ώστε όλοι να υποχρεωθούν να υλοποιήσουν το κείμενο. Η κυρία Πιλάρα Γιούσο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάννα Σέντερ, συγγνώμη. Ναι, ναι ε, νομίζω ότι ε, ε, σίγουρα, σίγουρα όλοι μας από κάπου μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να βρούμε θετικές λύσεις όσον αφορά την Ευρωβινέτα. Ευρωβινέτα προβλέπετε κάποια η μορφή αντιστάθμισης για τις πιο περιφερειακές χώρες. Επίσης τα πραγματικά προστιθέμενα κόστη τα έχετε λάβει υπόψη ή αποσπασμένη εργασία εργαζόμενοι. Ε, ε, ίσως, ε, ίσως αυτό μπορέσει να αποτελέσει μια καλή αρχή έτσι ώστε να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς κινητικότητας πάντα. Ε, επίσης, πώς θα ε, αποφύγουμε ε, να, γίνει όμοιρος τελικά ο αποσπασμένος εργαζόμενος και πώς μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Τέλος, ασφαλής χώρη στάθμευσης και αξιοπρεπής στέγη. Στην η είχε περιλάβει και το θέμα αυτό ήδη έτσι ώστε ε, να υπάρξουν τέτοιου είδους ε, ασφαλείς χώροι. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ε, ερωτών. Ευχαριστώ. Το πακέτο κινητικότητας που υποβάλλεται έχει 8 νομοθετήματα για τις οδικές μεταφορές. Έρχονται και άλλα για τις αναέρειες μεταφορές κτλ. και ιδίω για τις συνδυασμένες μεταφορές. Δεύτερο, οι πρώτες αντιδράσεις για το καμποτάζ των επιχειρήσεων τη εκλογική μου περιφέρεια είναι συντηρητικέ. Όλε οι επιχειρήσει αυτέ θεωρούν ότι ανοίγεται τελείω το καμποτάζ. Με ποιον τρόπο να του καθισχάσω του ανθρώπου αυτού. Σα ευχαριστώ, αγαπητέ και Κοχ. Κυρία Επίτροπε. Ε, ε, έχετε πολλές ερωτήσεις να απαντήσετε. Καμποτάζ, ευρωβινέτα και ούτω καθεξής. Έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, όλες οι ερωτήσεις σας είναι βεβαίως αξιόλογες και ενδιαφέρουσες και όλες αξίζουν μια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν είμαι βεβαίω ότι θα μπορέσω να σας ικανοποιήσω όλες και όλους, να σας δώσω δηλαδή πλήρε απαντήσεις. Σας παρακαλώ όμως να επανέλθετε και θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό για να εξηγήσουμε, να διευκρινίσουμε όλα τα σημεία του πακέτου. Να έρθω τώρα σε ορισμένε από τι ε, πιο γενικό, ε, γενικότερες ερωτήσει ή θέματα που ανέφερε και η Πρόεδρό σα. Πολλέ ερωτήσει αναφέρθηκαν στον χρόνο αναπαύσεως ή στου κατάλληλου χώρου στάθμευσης για του οδηγού. Οφείλω να ομολογήσω ότι υπενθυμίζουμε διαρκώ στι χώρε μέλη ότι πρέπει να διασφαλίσουν και σήμερα ακόμη οφείλουν να διασφαλίζουν ασφαλείς χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων για, τους, ε, για, χάρη των οδηγών. Και ε, η οδηγία προβλέπει στην λίστα των project που θα πρέπει να υποβληθούν για την συγχρηματοδότηση περιλαμβάνονται και ασφαλείς χώροι στάθμευσης. Αυτού του είδους τα έργα είναι κατάλληλα επίσης και για το blending και για project FC. Ασκήστε πίεση στις χώρες μέλη σας να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για να ε, εγγυθούν την ασφάλεια των οδηγών στους χώρους στάθμευσης. Εγώ θα σας είμαι ευγνώμων αν μπορέσετε να επανέλθετε και να μου πείτε πού ε, εντοπίζετε ανεπάρκειες και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε έξτρα ε, βοήθεια, οικονομική δηλαδή, για την κατασκευή των χώρων αυτών. Δεύτερο, ερώτημα που επανελήφθη ήταν σχετικά με την ψηφιοποίηση, τα ε, τέλη χρήσεως των δρόμων και ούτω καθεξής. Οι χώρες μέλη έχουν το δικαίωμα ακόμη να αποφασίσουν εάν θα επιβάλλουν διόδια ή όχι. Επομένως δεν είναι υποχρεωτικό. Αν αποφασίσουν ωστόσο να χρεώσουν διόδια, μετά από το 2027 θα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα υπολογισμού τη απόστασης και να περιλαμβάνει και τα εξωτερικά στοιχεία του κόστους. Δηλαδή δίνουμε 10 χρόνια σε όλους για να προσαρμοστούν, το οποίο εγγυάται την προβλεψιμότητα για τα ε, επενδυτικά έργα και για τους επενδυτές να γνωρίζουν τι τους περιμένει. Προσκαλούμε λοιπόν τους πάντες όσοι κάνουν λύσεις, όσοι προωθούν λύσεις ε, με ψηφιακό χαρακτήρα, να δημιουργήσουν και τις υποδομές για την προσαρμογή των μηχανισμών που θα χρησιμοποιήσουν. Γιατί πάλι distance-based, διότι η Ευρωβινιέτα όπως είναι σήμερα δεν περιλαμβάνει, δεν εντάσσει, δεν συμπεριλαμβάνει τα externality, δηλαδή τα εξωτερικά στοιχεία. Εμεί θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να τα περιλαμβάνει. Είναι ο μόνος τρόπος λοιπόν αυτός. Όσον αφορά την ισορροπημένη προσέγγιση του χρόνου 2018, θα είναι το έτος της πολυτροπικότητας, multimodality, θα ξανάρθουμε σε όλα τα θέματα. Πώς να συνδυάσουμε τους τρόπους καλύτερα και να διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα, πολυτροπικές λύσεις και ούτω καθεξής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψάχνουμε να βρούμε τους ελείποντες κρίκους, πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Να υπάρχει δηλαδή ένα ανεμπόδιστο ε, επίπεδο χωρίς κανένα, ε, κανένα σημείο ραφής χωρίς κανένα κενό, εν πάση περιπτώσει, σε όλη την Ευρώπη για την, για την ψηφιοποίηση. Χωρίς να είναι οι ίδιες οι επιβαρύνσεις σε κάθε χώρα μέλος. Αλλά θα χρησιμοποιούνται οι ίδιοι μηχανισμοί και τα ίδια πρότυπα. Και γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει μια νέα ευρωπαϊκή Δύση. διότι αυτή η κατακαιρματισμένη προσέγγιση δεν εξυπηρετεί τις διασυνοριακές υπηρεσίες, την προσφορά διασυνοριακών υπηρεσιών. Και η όλη υπόθεση της ενιαίας ε, αγοράς είναι να προσφέρει τις ε, προϋποθέσεις για διασυνοριακή προσφορά υπηρεσιών. Να υπάρχει λοιπόν ε, μια ενιαία θηρίδα στην οποία να μπορεί να απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος. Για πρώτη φορά θα έχουμε carrier business. Θα έχουμε και service subscription με κάποιον από τους παρόχους και αυτοί πλέον θα ασχολούνται ε, να υπάρξει σε όλο, ε, κίνηση σε όλη την ε, Ευρώπη. Δηλαδή πολλές υπηρεσίες που θα παρέχονται από έναν πάροχο. Θα αποτελέσει πρόκληση αυτό για πολλές χώρες, διότι συγκλονίζει συνθέμελα κάτι με το οποίο είχαν βολευτεί όλοι, έστω και αν δεν ήταν καλή, καλή η λύση. Αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι θα είναι πρόκληση αυτή, αλλά σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας να αναδιαμορφώσουμε τις μεταφορές μέχρι το 2030. Οι επιχειρήσεις ήδη επενδύουν σε διασυνδεδεμένες λύσεις, σε αυτόνομες λύσεις. Και αυτό είναι ένα αναγκαίο βήμα για να ε, μπορέσουν να γίνουν προσαρμογές αυτές. Σε ό,τι αφορά το γραφειοκρατικό άχθος, ακόμα και για μικρές επιχειρήσεις μεταφορών, θα δείτε και μπορούμε να σας δώσουμε και όλες τις αναλύσεις που έχουμε κάνει. 60%, 60 του ε, γραφειοκρατικού βάρους θα αυξηθεί. Μεγάλο νούμερο αυτό. Και με όλες αυτές τις ανταλλογές δεδομένων η έλεγχη στα σύνορα δεν θα χρειάζεται να κουβαλάν μαζί τους τρεις και τέσσερις βαλίτσες έγγραφα. Θα γίνεται με ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διοικήσεων. Και αυτή, αυτό το μητρό της ERU του Ευρωπαϊκού, το Ευρωπαϊκό Μητρό δηλαδή για τις επιχειρήσεις ε, οδικών μεταφορών θα έχει καταχώρηση και του οδηγού. Είναι τεράστια λοιπόν η απλοποίηση από την ε, πλευρά αυτή. Ελπίζω λοιπόν όμως βέβαια ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να σας τα εξηγήσω αυτά, δεν μου μένει πια πολύ χρόνος. Οι χώρες μέλη θα αποφασίσουν ποιες οδούς θα επιβαρύνουν με διόδια. Θα το επιβάλλει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή όμως το επιβάλλουν, επιβάλλουν τα τέλη αυτά. Δεν θα υπάρχουν πλέον 5 και 10 ε, διαφορετικά στίκερ που μετά θα πρέπει να τα αφαιρείτε με δυσκολία όταν θα χρειάζεται. Και ε, θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Και αυτή θα είναι και η υποδομή για τα φορτηγά, που γίνεται νομίζω 2023, ε, νομίζω, γίνεται υποχρεωτικό το σύστημα αυτο αυτοδιοδίων. Θα υπάρχει όμως τότε ήδη όλη η υποδομή. Έχουμε λοιπόν υπόψη μας ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και αυτά τα νούμερα βέβαια δεν μας ήρθαν έτσι. Ζητήσαμε από όλους τους παρόχους υπηρεσιών συστημάτων διοδίων πόσο χρόνο χρειάζεστε, ποιος είναι ο επόμενος κύκλος επενδύσεων. Και αυτοί μας έδωσαν τα νούμερα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη και ε, τους κύκλους απόσβεσης των υφισταμένων υποδομών τους Ευχαριστώ, κύριε κυρία Επίτροπε. Ε, μείνετε λίγο περισσότερο μαζί μας. Πάντως νομίζω ότι ε, θα πρέπει να σας συγχαρούμε ε, για, την, ε, ε, για τις απαντήσεις που μας δώσατε, για την παρουσία σας. Είναι το, το πακέτο κινητικότητας, ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και με μεγάλες συνέπειες, το είπατε και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ και που ανταποκριθήκατε σε όλα τα αιτήματά μας και φαντάζομαι ότι και ελπίζω ότι θα συνεχίσετε και στο μέλλον. Η Επίτροπος θα μείνει μαζί μας, αλλά θα ζητήσω μια σύντομη ε, διακοπή έτσι ώστε να σταματήσει η μετάδοση μέσω διαδικτύου και επίσης ε, να, εγκαταλείψουν, ε, να εγκαταλείψει το κοινό την αίθουσα γιατί θα συνεχίσουμε και κλεισμένων των θυρών. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αρμοδιότητα να παραμείνουν στην αίθουσα παρακαλώ να την εγκαταλείψουν. Οι βουλευτές να μείνουν βέβαια.